πρέπει να έρθουν εδώ και το κοινό που έρχεται από την άλλη αίθουσα. Or ίσως μπορώ και να αρχίσω εδώ που τα λέμε, γιατί έχουμε ένα-δυο θεματάκια πριν τους προσκεκλημένους μας. Πρώτα απ' όλα είχαμε στην άλλη αίθουσα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Περνάμε στο σημείο 2, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, δεν έχει προτείνει κανείς αλλαγές, εγκρίνεται. Καλώς. Ευχαριστούμε. Κάποιες ανακοινώσεις. Η πρώτη μου ανακοίνωση είναι ότι θέλω να σας θυμίσω ότι δυόμιση αρχίζουμε αύριο το απόγευμα. Τρίτη και Τετάρτη στις δυόμιση θα αρχίζουμε αντί για τις τρεις. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Link για να μπορούν Τρίτη και Τετάρτη να τελειώνουν ακριβώς στις 6.30 οι διερμηνείς. Τη Δευτέρα αρχίζουμε αργότερα για να έχει καιρό κόσμος να ταξιδέψει. Τώρα αύριο το μεσημέρι, να ξέρετε, υπάρχει μια συνάντηση με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πρόσφατη έκθεση ΟΗΕ και Παγκόσμιας Τράπεζας για την πρόληψη βίων συγκρούσεων. Αύριο, 12.45 λοιπόν, μέχρι τις 2 και στην αίθουσα PHS 5Β001. Μόνο στα αγγλικά, να ξέρετε. Και θα υπάρχουν και σάντουιτς. Σας ενημερώνω επίσης και για την επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Ασφάλειας της Γουατεμάλα, Άουρα Λετήθια Ντελεγουάριο. Θα ήθελε ο Υπουργό να συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής μας για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της ε, Γουατεμάλα κυρίως ε, την εθνική πολιτική για την ε, πολιτική απασχόλησης, αξιοπρεπούς απασχόλησης 2017-2032. Ήρθε κάπως αργά το έτοιμο, οπότε αυτό που είπαμε είναι ότι αύριο στο τέλος της συνεδρίασής μας ελπίζουμε να έχουμε ένα τέταρτο 20 λεπτά να συναντηθούμε μαζί της. Ελπίζω να είσαστε παρόντες κι εσείς. Σημείο 4. Ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσεις να μας κάνει. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, όχι. Ωραία. Οπότε περνάμε έτσι στο σημείο 5. Ακόμα όμως δεν έχουμε εδώ τους προσκεκλημένους μας. Από ό,τι μου είχαν πει, μόλις πριν από 5 λεπτά φεύγαν από την αίθουσα πρωτοκόλλου. Οπότε πούντι. Θα δούμε. Πάντως αύριο να ξέρετε ότι έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες. Στις 9, αύριο. Α, όχι, όχι, λάθος. 10 και 4 είναι η ψηφοφορία, 9 είναι οι συντονιστές. Μην μπερδευτούμε. Ωραία, με ιδιαίτερη χαρά. Μπαίνουμε στο σημείο 5, αγαπητοί συνάδελφοι, και πρόκειται για συζήτηση που θα έχουμε με τον πρόσφατα ορισμένο Γενικό Διευθυντή της, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τον κύριο Τέντρος. Είχα συναντηθεί μαζί του όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Αιθιοπίας όπου είχε κάνει τότε σημαντικές αλλαγές, βελτιώσεις στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας του τότε. Ε, ξελέχθη λοιπόν το Μάιο του 2017 Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας, πολύ σωστή στιγμή που σας συναντάμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο ε, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα προχωρήσει για να υλοποιήσει τους στόχους της χιλιετίας πώς θα καλύψει τα θέματα υγείας, ε, έκτακτες περιπτώσεις όπως ήταν η κρίση ε, έμπολα, τι θα γίνει με την υγεία των μητέρων και μένα να ξέρετε με ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερο το θέμα των καπνών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Υπήρξε μια έκθεσή σας πρόσφατα για τα καπνά, σωστά. Οπότε, δόκτωρα Τέτρος, Συγγνώμη που σας καθυστερήσαμε, οπότε έχετε το λόγο. Παρακαλώ και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και η Δόκτωρ Γιάκοπη είναι εδώ μαζί σας και εσείς καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, υπό διαφορετική ιδιότητα βέβαια αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Από πλευρά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας θέλουμε ε, τερική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πολύ χαίρομαι που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω και να απευθυνθώ σε εσά. Ειλικρινά χαίρομαι γι' αυτό. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανάπτυξης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να στηρίξει αναπτυσσόμενες χώρες να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν τους στόχους της χιλιετίας. Ο ΠΟΗ έχει δουλέψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και κοινά προγράμματα μεταξύ μας, όπως είναι η εταιρική σχέση που έχουμε και θα συνεχίσουμε σίγουρα και θα επεκταθούμε περισσότερο και στο θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα. Ξέρω ότι συζητάτε ένα νέο μηχανισμό προκειμένου να υπάρχει επαφή με την κοινωνία των πολιτών και ειλικρινά ελπίζω ότι ο μηχανισμός αυτός ο νέος θα δώσει τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι ιατρικές νοσηλευτικές ομάδες ώστε να υπάρχει εκπαίδευση και κατάρτιση παντού στον κόσμο. Εδώ και νέα μήνες ξεκίνησε ως Γενικός Διευθυντής στην ΠΟΕ και ήταν μια ιδιαίτερα εντατική και καρποφόρα περίοδος για μένα. Επικεντρωθήκαμε πρώτα απ' όλα στο να βάλουμε τις βάσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια. Να δούμε ποιοι θα είναι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ένα στρατηγικό σχέδιο με την αποστολή μας, προκειμένου να διατηρηθεί ο κόσμος ασφαλής και να βοηθήσουμε τους περισσότερο ευάλωτους. Το εκτελεστικό μας ε, Συμβουλίο τώρα έχει εγκρίνει το σχέδιο αυτό και στη Γενική Συνέλευση τον Μάιο περιμένουμε οι χώρες μέλη επίσημα να τον κρίνουν. Κανονικά παίρνει δύο χρόνια για να ετοιμάσει κανείς το επόμενο στρατηγικό σχέδιο. Εμείς όμως το κάναμε αυτό μέσα σε 8 μήνες. Δράσαμε γρήγορα γιατί είναι τεράστιες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και το κόστος της αναμονής είναι τεράστιο. Το σχέδιο στρατηγικής λοιπόν περιλαμβάνει τρεις φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια να έχουμε ένα δισεκατομμύριο ακόμα ανθρώπου οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εφημερία, να έχουμε καλύτερη προστασία από έκτακτες ε, περιστάσεις και ένα δισεκατομμύριο περισσότεροι άνθρωποι να περάσουν στην ευημερία. Έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε και για τους τρεις αυτούς στόχους. Θέλουμε οικουμενική κάλυψη σε όσο γίνεται υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή γι' αυτό έχουμε εισάγει μια νέα προσέγγιση σε περίπτωση εκτακτής ανάγκης όπου εμπλέκεται και το Συμβουλίο ε, του ΠΟΗ για όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης παγκοσμίω και το πώς ο ΠΟΗ αντιδρά. Έχουμε επίσης ετοιμάσει μια επιτροπή υψηλού επίπεδου για τις κολλητικές ασθένειες υπό το πρόεδρο της Ουρουάης. Θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν επίσης τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και εξακολουθούμε να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά την αντιμικροβιακή αντίσταση. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αλλάξουμε. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε μία διαδικασία προκειμένου να αλλάξει η ΠΟΗ και να δώσει περισσότερη σημασία στα ζητήματα τα οποία έχουν σημασία στις διάφορες χώρες. Επίσης, η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στις ηγετικές θέσεις της ΠΟΗ είναι μια υπόσχεση που είχα δώσει από πριν. Και για πρώτη φορά οι γυναίκες τώρα είναι παραπάνω από τους άντρες στις ηγετικές θέσεις. Και θέλουμε να την πετύχουμε σε όλα τα επίπεδα. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, φέτος έχουμε 100 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όμως είναι και 100 χρόνια από κάτι άλλο, το οποίο σκότωσε πολύ περισσότερους ανθρώπους από τον ίδιο τον πόλεμο και ήταν η επιδημία της Ισπανικής γρίπης, η οποία παραμένει η πιο θανατηφόρα επιδημία ανά τους αιώνες. Όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι και σήμερα μία επιδημία μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε χώρα, να πάσα στιγμή και να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουμε, γιατί είμαστε ακόμα ευάλωτοι. Ευτυχώς ε, δεν έχουμε δει τέτοια επιδημία έκτοτε, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να συμβεί. Και εξακολουθεί ο κόσμος να είναι ευάλωτος. Μερικές φορές είναι θέμα τύχης AIDS για παράδειγμα που ξεκίνησε το 2003 πάρα πολύ Το επικίνδυνο HJ1 επίσης το στέλεχος. Το H1N1 επίσης η πανδημία αυτή του 2009 ε, μεταδόθηκε πάρα πολύ εύκολα μεταξύ του κόσμου, αλλά ευτυχώς σε ήπια μορφή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και βέβαια η τεράστια κρίση ήταν ο έμπολα που έπληξε τις χώρες της Δυτικής Αφρικής και έπληξε και ολόκληρη την ασφάλεια της περιοχής. Πέρα από το ανθρώπινο κόστος, επίσης ο ιός του έμπολα είχε και οικονομικές επιπτώσεις. Το IMF μείωσε τις προσδοκίες του για τις τρεις αυτές χώρες που επλήγησαν. Η ανεργία αυξήθηκε, η δημοσιονομική κατάσταση επιδεινώθηκε. Μας έδωσε μαθήματα όμως ο ιός του έμπολα. Ότι ένα ευάλωτο σύστημα σε μια χώρα μπορεί να δημιουργήσει μια παγκόσμια καταστροφή στην υγεία. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε τόσο ισχυροί όσο ο πιο αδύναμος κρίκος μας τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι κατάλληλα. Αν δεν είναι ή αν δεν εργάζονται ικανοποιητικά το νοσηλευτικό προσωπικό, είτε επειδή δεν πληρώνεται αρκετά, επειδή δεν έχει καταρτιστεί αρκετά ή επειδή ένας κρίκος στην αλυσίδα λείπει, η καταστροφή παραμονεύει στη παραμονεύει η μεγαλύτερη απειλή στην παγκόσμια ασφάλεια είναι ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας η υγεία, η ασφάλεια αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η πραγματικότητα είναι ότι ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στη φτώχεια επειδή αναγκάζονται να πληρώνουν για την υγεία τους από τα δικιά τους την τσέπη αν δεν έχουν βοήθεια, υπηρεσίε υγεία κοντά στα σπίτια τους ή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, μπορεί να μην ληφθεί υπόψη το πρώτο δείγμα έκρηξη μια νέας επιδημίας. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί μόνο τότε μπορούμε να σταματήσουμε μια πανδημία στην αρχή της. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις εμπειρίες που έχουμε από το παρελθόν και να ξέρουμε ότι είναι ευάλωτε όλε οι χώρε, όλα τα επίπεδα. Και όλε οι χώρε, όλοι οι λαοί μπορούν να κάνουν περισσότερα με του πόρου που διαθέτουν. Αυτό σημαίνει ότι για τι περισσότερε χώρε ο μοναδικός φραγμός που υπάρχει είναι πολιτική βούληση. Γιατί τελικά η οικονομική κάλυψη είναι θέμα πολιτικής επιλογής και τίποτα άλλο. Πολλέ χώρες, ιδίω εδώ στην Ευρώπη, την έκαναν αυτή την επιλογή για την οικονομική κάλυψη. Η Κίνα, η Ρουάντα, η Ταϊλάνδη και άλλες χώρες προχωρούν στην επιλογή αυτή. Ήμουνα στην Κένια πρόσφατα, όπου ο πρόεδρος είπε ότι θα αποτελέσει έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της οικονομίας για το δεύτερο ήμιση της θητείας του αυτή ακριβώς η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και η Ινδία επίση είπε 12% αύξηση στον προπολογισμό για την υγεία, που σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να καλυφθούν και θα δημιουργηθούν 150.000 κέντρα Όταν ήμουν εκεί, όταν συζητήσαμε για το δικό του το πρόγραμμα με τους Ναμπαχάρα, είδα ότι υπάρχει ενέργεια και διάθεση όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, αλλά και στους ίδιους τους νοσηλευτές, το νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί υπάρχει αυτή η φιλοδοξία για την οικουμενική κάλυψη. Όμως τα ωφέλη δεν είναι μόνο για την υγεία. Οι επιδημίες, όπως είπαμε, μπορούν να πλήξουν την οικονομία. Συνεπώς, η οικουμενική κάλυψη μπορεί να βοηθήσει την οικονομία των χωρών. Να βοηθήσει δηλαδή να υπάρξει και περισσότερη οικονομική αντοχή. τα παιδιά όταν ενηλικιώνονται γίνονται παραγωγικά στοιχεία της κοινωνίας. Όταν οι γυναίκες δεν πεθαίνουν στη γέννα, μπορούν να ασχοληθούν με τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους. Όταν δεν υπάρχει ρήπανση, μόλυνση, επικίνδυνα προϊόντα, υπάρχει ευημερία. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε πού, ούτε πότε θα ξεσπάσει η νέα επιδημία. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι θα πληρωθεί τεράστιο τίμημα και σε ανθρώπινη ζωή αλλά και οικονομικά. Μπορεί να υπάρξει και πολιτική αστάθεια. Όπως είπα, το κλειδί είναι να τον αγνωρίσουμε αυτό, να έχουμε την οικουμενική κάλυψη, γιατί η οικουμενική κάλυψη για την υγεία και η οικονομία είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, όπως είπαμε. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε τον ιστό των συστημάτων υγείας παντού. Εξού και η ΠΟΕ δουλεύει παντού στον κόσμο για να ενισχύσει τέτοια συστήματα, για να ενισχυθεί η κάλυψη υγείας, η πρόληψη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Είπαμε, υπάρχει τεχνική πτυχή, υπάρχει και πολιτική πτυχή. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή η πολιτική για αυτήν την οικουμενική κάλυψη. 7 Απριλίου ξεκινάμε μια εκστρατεία διετή για να υπάρξει νέα πολιτική δέσμευση υπέρ της οικουμενικής κάλυψης. Και στην Γενική Συνέλευση τον Μάιο θα ζητήσουμε από όλες τις χώρες να αναλάβουν τρία βήματα προκειμένου να πετύχουν αυτήν την οικουμενική κάλυψη και να την κάνουν πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πολύ σημαντικό εταίρο μας αυτή την προσπάθεια οικουμενικής κάλυψης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εταίρων μας στηρίζεται το σύστημά μας αυτό σε 35 χώρες. Και όπως είπα στην αρχή, έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και πρέπει να έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες γιατί οι προκλήσεις είναι τεράστιες για να έχουμε χαμηλούς στόχους. Αν όμως θέλουμε να πετύχουμε το όραμά μας για μια δίκαια υγεία, οικουμενική κάλυψη, χρειαζόμαστε τη δικιά σας τη στήριξη γιατί τελικά οι δικές σας οι επενδύσεις βελτιώνουν και την υγεία των ανθρώπων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργούν και μια πιο ασφαλή Ευρώπη, έναν πιο ασφαλή κόσμο, αποφεύγοντας ε, Η Επιτροπή σας επίσης μπορεί να παίξει ένα ρόλο κλειδί τα επόμενα χρόνια. Στη σημερινή συζήτηση που γίνεται για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για τα επόμενα 7 χρόνια, πρέπει να θυμόμαστε ότι η υγεία, η ευημερία είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη παντού στον κόσμο και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πραγματικής αλληλεγγύης. Αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει οικονομία και ούτε μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα μαζί. Αυτό όμως που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι εμείς είμαστε τόσο δυνατοί όσο πιο αδύναμος κρίκος μας. Γι' αυτό και η αλληλεγγύη είναι το στοιχείο κλειδί. Το μόνο όριο, ο μόνος περιορισμός είναι το μέγεθος των φιλοδεξιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much. I was very pleased when... Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, είχαμε αυτή την επιτροπή, γιατί αυτά που είπατε πραγματικά ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Μουσική στα αυτιά μας τα έλεγα. Ε, ως ε, επιτροπή μετά την κρίση του έμπολα μπορέσαμε να διαπιστώσουμε μόνοι μας τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρεται όπου υπήρχε σύστημα υγείας, αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Σε άλλα που δεν υπήρχε σύστημα υγείας, θα μπορούσε να προκύψει πραγματικά μια οικουμενική καταστροφή. Και δαπανίσαμε δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Ε, μάλιστα θα έχουμε μια αποστολή στη Γουινέα για να δούμε επιτόπου τι ακριβώς έχει προκύψει γιατί θυμάμαι ένα από τα μηνύματα ήταν ε, αυτά που ε, αφορούσαν τα παιδιά να σώσουμε τα παιδιά. Και αν είχαμε επενδύσει σε αυτέ τι χώρε σε σύστημα υγεία, δεν θα υπήρχε πρόβλημα εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα το σύστημα υγεία είναι καθοριστική σημασία και είναι και θέμα πολιτική επιλογή. Στη δική μου τη χώρα έχουμε το Εθνικό Σύστημα Υγεία και το φτιάξαμε το 1947. όχι όταν ήμασταν πλούσια, αλλά αμέσω μετά τον πόλεμο, όπου ήμασταν τραγικά χρεωμένοι, μεγάλη κρίση τότε, υπήρχε έλλειψη ε, πρώτων υλών, αλλά τότε λάβαμε την απόφαση ότι η υγεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τη τελική ανάλυση η υγεία φέρνει οικονομική ανάκαμψη ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Γκερέρο είναι ο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται χρόνο να βάλετε τα ακουστικά σας. Περιμένω. Έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για τη δουλειά που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ε, μας παρουσιάσατε κάποιες από τις ε, βασικές γραμμές και όπως μόλις είπε η Πρόεδρος Επιτροπής, οι συζητήσεις για τη σχέση μεταξύ πολιτικές, ε, πολιτικών ανάπτυξης ε, και υγείας ε, και το πώς εντάσσονται σε αυτές τις πολιτικές είναι θέμα το οποίο μας απασχολεί μονίμως εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης και ταυτόχρονα η απάντησή μας στην κρίση του έμπολα ήταν συνεχής και ταυτόχρονα πολύ συγκεκριμένη και έτσι ορίσαμε και έναν ειδικό εισηγητή για τον έμπολα ο κύριος Γκέρενς ε, ανέλαβε τα καθήκοντα μέλος της Επιτροπής. Και θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση ε, απλή σχετικά. Εγώ ήμουν εισηγητής για την ανθρωπιστική δράση και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις ανθρωπιστικές κρίσεις κρίσεις οι οποίες ξεσπούν αυθόρμητα, όπως για παράδειγμα οι κρίσεις μακράς διαρκείας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κάνει ο ΠΟΗ σε τέτοιες κρίσεις, τι δουλειά κάνει και με ποιες άλλες ε, οργανώσεις και οργανισμούς, τη UNICEF, ε, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ή κάποια άλλη οργάνωση, συνεργάζεστε επί τόπου στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης για την αντιμετώπιση των διάφορων κρίσεων που σοβούν τον κόσμο. Και επίσης ε, και ένα τελικό σχόλιο για την αδικία να αποκαλείται ισπανική γρήπη αυτό το οποίο συνέβη πριν από 100 χρόνια, γιατί όπως ξέρει όλος ο κόσμος, οι καταβολές της δεν ήταν στην Ισπανία. Είναι ιστορική αδικία αυτή το να ονομάζεται αυτή η πανδημία ισπανική γρήπη. Okay, thank you. Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς στηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, τα οποία έχουν προβλήματα με τις ε, επιδημίες ε. και επίσης αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρεται ικανοποιητική περίθαλψη στους πολίτες. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας ε, τότε που είχαμε, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση του έμπολα, διαπιστώσαμε το εξής, ότι οι χώρες με περιορισμένη ιατρική περιθαλψή, οι χώρες αυτές επλήγησαν περισσότερο. Δεν θέλω να το αξιολογήσω απαραίτητα, αλλά το τεκμηριώνουν τα στοιχεία είχαν λιγότερους γιατρούς, ε, λιγότερο ιατρικό προσωπικό. Δυστυχώς λοιπόν το γεγονός αυτό οδήγησε στο ότι επίσης η ιατρική περίθαλψη περιορίζεται στις πρωτεύουσες αυτών των κρατών. Υπάρχουν ε, γιατροί οι οποίοι θα έπρεπε να προσφέρουν ε, περίθαλψη ε, και πέρα και μακριά από την πρωτεύουσα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο απαραίτητα. Ε, δυστυχώς ε, ε, όσοι δεν ζουν στην περιφέρεια, στην πρωτεύουσα, δεν έχουν ικανοποιητική ιατρική περίθαλψη. Πόσο μάλλον όταν ξεσπάει επιδημία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ερωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε ότι κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά πολλά χρήματα για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Οι επιπτώσεις, ακριβώς όταν πρόκειται για την ε, ιατρική περίθαλψη, ε, οι επιπτώσεις, οι, οι θετικές συνέπειες δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακέ. Εσείς έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να μπορούν να προσφέρουν καλύτερη ιατρική περίθαλψη, περίθαλψη υγείας, δηλαδή να προσφέρεται περίθαλψη όχι μόνο στις πρωτεύουσες αλλά και στα μικρά χωριά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νόιζα. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ευχαριστώ πολύ και εσάς ε, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εσείς αλλά και η Πρόεδρος μας πολύ σωστά δείξατε ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε με τις χώρες εκείνες που έχουν ε, τροτά συστήματα υγείας. Τρομάξαμε με την ε, κρίση του Ιουέμπολα, αλλά εκτός από τη Λιβερία, τη Γουινέα, υπάρχουν και άλλα κράτη ε, που έχουν τροτά συστήματα υγείας. Δεν ξέρω μάλιστα αν μετά αυτήν την κρίση με τον ιό έμπολα κατά πόσον ε, πράγματι μάθαμε το μάθημά μας. Γιατί εγώ πήγα δύο φορές ε, στη Σχέρα Λεόνε και σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε αυτά τα ταξίδια δεν διαπίστωσα να έχει βελτιωθεί η περίθαλψη υγείας. Πολλές ΜΚΟ εγκατέλειψαν αυτές τις χώρες, τώρα πια αυτές οι χώρες ε, ε, σχεδόν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, προκλήσεις. Η δική μου ερώτηση είναι τι είδου επιρροή μπορεί να ασκήσει ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας έτσι ώστε σε αυτές τις τρεις χώρες που ανέφεραν δεικτικά να επικρατήσει μια σταθεροποίηση. Το τρίτο θέμα αφορά εμάς και εκείνα τα οποία πρέπει να πράξουμε στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Αν δούμε λιγάκι τώρα το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που συζητείται και βλέπουμε ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο ε, θα διαχωρίζεται από θέματα μετανάστευσης ε, και πολιτικής μετανάστευσης. Ε, η αντιμετώπιση της φτώχειας ε, φοβάμαι ότι είναι απολύτως απαραίτητη για να υπάρχει και ικανοποιητική περίθαλψη υγεία. Το ίδιο ισχύει και η την υγεία. Δυστυχώς όμω δεν φαίνεται να συμμερίζονται και άλλοι την άποψή μου. Ε, θέλω το 2014 να μην ε, επαναληφθεί. Δεν θέλω για άλλη μια φορά να σοκαριστούμε επειδή εντάξει θα έχει ξεσπάσει επιδημία. Οι χώρες, ε, όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες να είναι πρόθυμες να διαθέσουν ξαφνικά κάποια κονδύλια, αλλά δεν θα υπάρχει συνέχεια. Αυτό δεν μπορεί να φτάνει από μόνο του. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα μέτρα εκείνα που προτείνετε έτσι ώστε να υπάρξουν θετικές συνέπειες στις ε, θυγόμενες χώρες και να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά που μας είπατε και έχω να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως ε, πρώτα απ' όλα να σας ε, παραπέμψω σε δύο συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία ε, προετοιμάζει αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. στις ε, επιτροπές μας ε, εργαζόμαστε πάνω σε μια έκθεση για ένα πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την υγεία και αφορά και ένα πολύ μεγάλο θέμα που θίξατε εσείς, δηλαδή την αντιμικροβιακή αντοχή. Αυτό είναι το πρώτο έγγραφο. Και το δεύτερο ε, τέτη υποβλήθηκε το Δεκέμβρη ή εγκρίθηκε από την ΑΚΕ το Δεκέμβρη και εκεί προβλέπεται καλύτερη πρόσβαση ε, σε θέματα ιατρικής ε, περίθαλψης και αυτό για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι μολυσματικές ασθένειες. Ίσως ε, λοιπόν αυτά να είναι κίνητρα που να είναι σημαντικά και για τη δική σας τη δουλειά. Και τώρα θέλω να περάσω κι εγώ σε δύο ερωτήσεις που έχω να σας υποβάλω. Όσον αφορά στο πρόγραμμα το οποίο εφήξατε, θα ήθελα να σας ερωτήσω πώς ακριβώς ε, το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εφαρμόστηκε στην πράξη, αν ε, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του και ε, σε ποιους τομείς διαπιστώσατε να υπάρχουν ελλείψεις τις οποίες θα πρέπει να περάσετε στο νέο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κέγγε. Σας ε, ευχαριστώ πολύ Λίντα και ευχαριστώ πολύ και τον ε, Δόκτωρα Τέντρος ε, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να οργανώσουμε από κοινού μια πρωτοβουλία. Γι' αυτό λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και στην Επιτροπή μας. θα πάω λίγο πίσω για να σας εξηγήσω και λιγάκι πώς ε, σήμερα προσπαθούμε να αλλάξουμε λιγάκι και την προσέγγιση, τη γενικότερη κατεύθυνση. Όμως, δυστυχώς, ε, ακόμα έχουμε να διανύσουμε μεγάλο δρόμο. Τη δεκαετία του 70 είχαμε ε, ένα σύνθημα που έλεγε μέχρι το 2000 υγεία για όλους. Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο, γιατί το πρόγραμμα αυτό βασιζόταν στην ισότητα. Ενώ μετά από κάποια χρόνια διαπιστώσαμε ότι η σωστή λέξη δεν ήταν η λέξη ισότητα, Γκουαλιάντσα, αλλά ίση αντιμετώπιση, εκουητά. στην περιοχή όπου ζει κανεί ε, θα πρέπει να έχει και την ίδια πρόταση, με αυτή την έννοια της ε, ίσης προσέγγισης και τοποθέτησης. Ε, το 2000 ξεχάσαμε ένα συγκεκριμένο πράγμα, να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ως εκ τούτου η υγεία και όλες αυτές οι προτάσεις ε, που καταθέτουμε δεν θα πρέπει να παραμένουν μόνο στον τομέα της υγείας. Επάνω από αυτές τις χώρες που θίγουμε, όταν μιλάμε για την υγεία, αυτομάτως ε, η υγεία είναι άμεσα συνδεμένη και με την ε, χερσαία και την οδική υποδομή. Δηλαδή, εκεί όπου στις ε, ε, περιφέρειες υπάρχουν κάποια κέντρα, αν δεν μπορεί κανείς να πάει, να μεταβεί, αυτό αποβαίνει μοιραίο. ω εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να φτιάχνει κανείς ένα νοσοκομείο χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την γύρω-γύρω υποδομή. Η υποδομή είναι καθοριστική σημασία. Αυτό σημαίνει, συμβαίνει και με το περιβάλλον. Ε, αυτό συνέβη με τον έμπολα. Παραδείγματο χάνει η διαχείριση των αποβλήτων, η καθαριότητα κοινότητα εκεί που ζουν οι άνθρωποι. Αν όλα αυτά δεν ληφθούν υπόψη, τότε αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση, οποιαδήποτε λύση είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να διευρύνουμε την προσέγγιση μας και να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες τομείς για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Όσον αφορά τώρα την εμπειρία με τον έμπολα, εγώ πήγα στη Γουινέα και εκεί είδα και τις ε, προσπάθειες που καταβάλει η τοπική κυβέρνηση. Ξεκίνησαν να βελτιώνουν το σύστημα της υγιεινής και αυτό όχι μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία αλλά και σε μικρά κέντρα θέλουν να δώσουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να μπορέσουν να ε, έχουν πρόσβαση σε ένα γιατρό. Πρέπει λοιπόν αυτές οι μεταρρυθμίσεις να ενταθούν σε περισσότερες περιοχές ε, και τα κέντρα της τελειότητας, τα περιφερειακά. Γιατί αν δεν υπάρχει ένα περιφερειακό κέντρο το οποίο να μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για όποιον ε, αντιμετωπίζει, έρχεται αντιμέτωπο με μια επιδημία, αν δεν υπάρχει αυτό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Με τον έμπολα, ακριβώ αυτό ε, αντιμετωπίσαμε, ότι δεν υπήρχαν κέντρα περιφερειακά για να σώσουν του ανθρώπου. Ω εκ τούτου πρέπει να υπάρχει μεταρρύθμιση των συνθηκών υγιεινή, ε, ένα σύστημα εκπαίδευση επιτόπου, να υπάρχουν περισσότεροι γιατροί, νοσοκόμε, όλα αυτά επιτόπου. Και αυτά ξεκινάνε από την εκπαίδευση. Να υπάρχει και πρόσβαση πρόσβαση στα φάρμακα. Ε, θέλω να απογραμμίσω το εξή, ότι όταν γίνεται λόγος ε, για πρόσβαση στα φάρμακα στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος υγείας, πάρα πολλές χώρες στην Αφρική έχουν ε, σύγχρονη ιατρική αλλά και παραδοσιακή ιατρική. Σε ορισμένε χώρε κατέστηνατόν να, εν, να ενσωματωθούν αυτά τα δύο ήταν πολύ σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό αποφεύγει κανεί το να ε, χάνονται κάποιοι ασθενείς ε, γιατί αυτοί ε, παίρνουν φάρμακα που δεν είναι αναγνωρισμένα και δεν έχουν καμία θετική δράση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατά πόσον έχει λάβει υπόψη του όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, να εντάσσονται στην προσέγγιση πάρα πολλοί τομείς. Γιατί όσον αφορά το θέμα της υγείας, αν δεν λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον στο οποίο ζει κανείς, η υποδομή που είναι καθοριστική σημασία, ε, τότε ε, τα χρήματα τα οποία δίδονται στις ε, περιφέρειες θα πρέπει ακριβώς να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες. Κύριε Τέντρος, είχατε πολλές ερωτήσεις, κάποιες αρκετά διεξοδικές, αλλά αυτό νομίζω καταδεικνύει ότι οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά και τρεις από αυτούς ε, θα πάνε στη Γουινέα σε μερικές εβδομάδες. Επομένως, ε, περιμένουμε να δούμε και τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε από τον ιό έμπολα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απαντήσω τις ερωτήσεις ε, ακολουθώντας την ίδια σειρά. Ανάπτυξη και υγεία είναι αλληλένδετα, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βεβαίως ε, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, η υγεία είναι θέμα δικαιωμάτων ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και επίσης είναι και μέσο για την ανάπτυξη και την ευημερία. Επομένως είναι δύο σε ένα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και τα δύο σε θέματα πολιτικής Ιδίω όταν αναφερόμαστε στην υγεία για όλους ή την οικουμενική κάλυψη υγείας. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφής η την οικουμενικη καλυψη υγεια πρεπει λοιπον να ειναι σαφης η σχεση με την ανάπτυξη, αλλά ανεξάρτητα με τη σχέση που έχει η υγεία με την ανάπτυξη, είναι θέμα δικαιωμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι σαφές για σας και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Τώρα, για τις σχέσεις που έχουμε με άλλους οργανισμούς, ιδίως ε, ε, μετά από την εμπειρία με τον ιό έμπολα, ε, ήδη συμμετέχουμε σε πολλές ε, επιδημίες, αλλά ε, εμείς γνωρίζουμε περισσότερα όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον, από τον έλεγχο, όπως με τον ιό έμπολα. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε και κάπου αλλού έμπολα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά δράσαμε γρήγορα. Ο ΠΟΗ όμως δεν δραστηριοποιείται μόνος του. Συντώνησε όμως την όλη διαδικασία. Ε, μεταφέραμε ε, κονδύλια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ε, οργανώθηκε κυβέρνηση, συμμετείχαν και οι άλλοι, η MSF, η UNICEF, πολλές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε και έτσι πολύ γρήγορα καταφέραμε να επιτεθούμε στο πρόβλημα και να το θέσουμε υπό έλεγχο. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Επανόλη στη Μαδαγασκάρ. Δεν ξέρω αν το, το ήξερε όλο ο κόσμο. Σε κάποιε περιοχέ το γνωρίζουν. Αλλά ελέγχθηκε χωρί να τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή. Το γεγονό, ο τρόπο όμω που ξεκίνησε ήταν ε, επικίνδυνο. Υπήρχαν τρει συνδυασμοί οι οποίοι είναι θανάσιμοι. Ο πρώτο συνδυασμό, ο πρώτο παράγων ήταν ότι ξεκίνησε νωρίτερα από την αναμενόμενη περίοδο που περιμένουμε την εμφάνισή του. Ήταν δηλαδή σαν να μας εξέπληξε. Το δεύτερο ήταν ότι έπληξε μη ενδυμικές περιοχές πέραν των περιοχών στις οποίες ενδυμεί. Και τρίτον ήταν πνευμονική. Αυτή τη φορά χτύπησε στους πνεύμονες και αυτό είναι μοιραίο. Ο συνδυασμός των τριών είναι πολύ επικίνδυνος και μάλιστα το γεγονός ότι μας κατάλαβε εξαπίνει στο πιο συγκεκριμένο. Ε, ξεκίνησε τον Αύγουστο και μέχρι τον Νοέμβριο το είχαμε ελέγξει. Δεν πέρασε καν τα σύνορα. Και το τρίτο ήταν ο ιός Μάλμπεργκ ο οποίος ξεκίνησε στην Ουγκάντα, κατάφερε να περάσει και στην Κένια, είχαμε ένα περιστατικό, αλλά και αυτό το ελέγξαμε. Και αυτό διότι υπήρξε ταχεία ανταπόκριση όχι μόνο από τον Μπόι, αλλά και από τους εταίρους του. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όμως είναι αυτός ο οποίος συντονίζει, έχει το συντονιστικό ρόλο και αυτή τη στιγμή συντονίζει όλα τα θέματα υγείας όποτε υπάρχει ε, εξέσπασμα επιδημίας. Υπάρχει λοιπόν ένα καλύτερο σύστημα, χάρη στη μεταρρύθμιση που έκανε ο ΠΟΗ, και υπάρχει καλύτερη απάντηση, αλλά φυσικά ε, η αδυναμία μας ακόμα δεν έχει μειωθεί ουσιαστικά. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα συστήματα υγείας μας, κυρίως σε επίπεδο χώρας, προκειμένου να υπάρχει ε, εύρωστη και πολύ ισχυρή απάντηση. Εν δεν θα μας βοηθήσει η στήριξη έξωθεν, να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα, αλλά οι δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο χώρας είναι αυτές οι οποίες θα μας βοηθήσουν. Γι' αυτό και στην παρέμβασή μου είπα ότι είμαστε ισχυροί όσο ο αδύναμος ε, κρίκος. Και φυσικά ε, η λύση είναι να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας των πιο αδυνάμων ώστε να προστατεύονται όλοι. Μέχρι να προστατεύονται όλοι δεν θα είναι κανείς ασφαλής. Αυτό είναι το όλο σκεπτικό. Και αυτό ισχύει διότι ο κόσμος γίνεται όλο και μικρότερος και μέσα σε λίγες ώρες ένας ιός μπορεί να εξαπλωθεί πέραν των συνόρων και να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να επενδύσουμε στην πρώτη γραμμή, στις χώρες στις οποίες υπάρχει αδυναμία στα συστήματα υγείας, πρωτίστως. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και παρεπτόντως αυτό έχει σχέση και μία με μία από τις ερωτήσεις, είναι αν όντως αντλήσαμε διδάγματα. Και ναι και όχι. Ναι, διότι κάναμε μια απόπειρα να μεταρρυθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, κινούμαστε και βλέπουμε ότι έχουμε καλύτερη ανταπόκριση. Σας μίλησα για τις τρεις χώρες τις οποίες καταφέραμε να ε, διαχειριστούμε τις επιδημίες γρήγορα. Αλλά ταυτόχρονα και όχι, δεν νομίζω ότι αντιλήσαμε σωστά τα διδάγματά μας, γιατί υπάρχει και αυτός ο κύκλος του πανικού και της αμέλειας. Όταν ε, πανικοβάλλεται κανείς, επενδύει πάρα πολλά, ακόμα και δισεκατομμύρια για παράδειγμα στον ιό έμπολα. Ένα κλάσμα αυτών θα αρκούσαν εάν τα είχαμε επενδύσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Παρεπιπτόντως δεν επισκευάζει κανεί το σπίτι του όταν ε, την περίοδο των ε, βροχών, το επισκευάζει νωρίτερα, πριν ξεκινήσουν οι βροχέ. Αλλά όταν υπάρχει βροχή και το σπίτι έχει πλημμυρίσει, τότε μα πιάνει ο πανικό και επενδύουμε πολλά. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, δεν επενδύουμε. Για παράδειγμα, το Ταμείο Εκτάκτου Ανάγκης, ε, το οποίο συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη του ΠΟΗ και ε, συστήθηκε, ελάχιστες χώρες το χρηματοδοτούν. Και ε, αυτή τη στιγμή εξαντλείται η χρηματοδότηση για αυτό το Ταμείο Επίγουσας Ανάγκης, διότι βρισκόμαστε στην περίοδο της αμέλειας. Τα πράγματα φαίνεται να βαίνουν καλώς, φαίνεται να είναι σταθερά και επομένω δεν προσπαθούμε και να επενδύσουμε. Και αυτό προσπαθώ να πω, αυτό είναι το μήνυμά μου, ότι η στιγμή να επενδύσουμε είναι τώρα που βλέπουμε τα πράγματα να βαίνουν καλώς, όχι όταν προκύψει το πρόβλημα. Επομένω δεν έχουμε αντλήσει τα διδάγματά μα γιατί βλέπετε το Ταμείο Επίγουσα ανάγκη. το οποίο μα βοήθησε να κινηθούμε γρήγορα στη Μαδαγασκάρη, μα βοήθησε να κινηθούμε γρήγορα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καταφέραμε να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και στην Ουγκάντα και στην Ιεμένη και στη Συρία. Αλλά εξαντλούνται τα αποθέματα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιληφθούμε. Δεν έχουμε αντλήσει εν μέρη τα διδάγματά μας. Κάποια πράγματα τα μάθαμε, κάποια άλλα όχι. Μετά, ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών, ιδίω ε, με το ιατρικό προσωπικό, κυρίως χώρες οι οποίες πλήττονται οικονομικά, αυτά που λέει ο αξιότιμος βουλευτής ε, είναι σωστό. Οι περιοχές ε, του Άστεως έχουν καλύτερη κάλυψη επαγγελματιών, είτε είναι ιατροί, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Οι περιοχές της Υπέθρου δεν έχουν τόσο πολύ καλή κάλυψη. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, ο ΠΟΗ προσπαθεί να βοηθήσει χώρε να ε, προτείνουν μηχανισμού για δημιουργία κινήτρων για αυτού οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να μεταβούν στην Ήπεθρο. Η άλλη λύση είναι η εξή. Ποια, τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί τη συγκέντρωση των γιατρών στις αστικές περιοχές. Η έλλειψη ε, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν και στην εκπαίδευσή τους. Όταν λέω λοιπόν να επενδύσουμε στα συστήματα υγείας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στο νέο Πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, η συμβουλή μας ως ΠΟΗ είναι να επενδύσουμε στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας και ένα στοιχείο εξ αυτών είναι η ανθρώπινη πόρη. Αν υπάρχουν ελλείψεις ε, και καλυφθούν, τότε η κάλυψη των αστικών περιοχών και τις περιοχές του υπαίθρου θα είναι καλύτερη. Γιατί η προσφορά και η ζήτηση είναι αυτές οι οποίες ε, οδηγούν σε συγκέντρωση των λίγων γιατρών που διαθέτουμε στις αστικές περιοχές και δεν έχουμε κανένα να στείλουμε στην Ήπεθρο. αυτό είναι πάλι συστημικό πρόβλημα. Τώρα, όταν αναφερόμαστε σε ανθεκτικότητα σε επιδημίες, δεν είναι οι παράγωγες ε, υπηρεσίες ε, και τα πιο δευτερεύοντα νοσοκομεία τα οποία θα δώσουν τη μάχη για να αντιμετωπίσουμε την επιδομία νωρίτερα. Ίσα ίσα είναι τα, τα πρωταρχικά, τα κύρια νοσοκομεία και σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε. Και όπως ε, είπε πολύ σωστά ένας από εσά, επένδυση στα ουσιώδη είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όταν αναφέρομαι στα ουσιώδη, αναφέρομαι στη βασική ιατρική κάλυψη, ε, στην πρόληψη των νόσων. Και πρέπει να ξαναπάμε στα βασικά. Παρεμπιπτόντως, ένας από εσά αναφέρθηκε στο κίνημα του δεκαετία δεκαετίας του 70 που ξεκίνησε στο Αλμάντι και πράγματι ε, γιορτάσαμε την 40η επέτειο. Η βασική λοιπόν ιατρική ε, περίθαλψη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του κινήματος της οικουμενικής κάλυψης των συστημάτων υγείας. Σημαίνει ότι θα προωθήσουμε την υγεία και την πρόληψη που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και μεταδιδόμενες και μη μεταδιδόμενες ασθένειες. Αλλά η επένδυση στα βασικά είναι πάρα πολύ χαμηλή αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα βρίσκεται στο επίκεντρο βασική κάλυψη υγείας και όχι μόνο στις αστικές περιοχές αλλά και στις περιοχές της υπαίθρου. Αν επενδύσουμε στις περιοχές της υπαίθρου είναι εύκολο να καλύψουμε και τις ανάγκες και να έχουμε και ένα καλύτερο σύστημα. Τώρα, τι μπορούμε να μάθουμε από τις επενδύσεις που κάναμε στο παρελθόν και ε, τώρα. Ξέρω ότι υπήρχε ε, μεγάλη κάλυψη για τη φωματίωση, για το AIDS, υπήρχαν προγράμματα και εκστρατείε. Οι επενδύσει όμως για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα είμαι ευγνώμων σε όλους του εταίρους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επενδύουν στην ε, φυματίωση, στην ελονοσία, στο νιό του AIDS ε, αλλά ε, είναι εξίσου σημαντικά και τα συστήματα υγείας, η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, γιατί βοηθά το σύστημα να συνεχίσει να παλεύει. Όταν αναφερόμαστε σε επενδύσει σε συστήματα υγείας και ενίσχυση των ε, συστημάτων υγείας, επενδύουμε στο μέλλον. Ακόμα και τώρα λοιπόν, το να υπάρχουν επενδύσεις στα προγράμματα και επενδύσεις για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε δυνατότητες για τα συστήματα υγείας για δύο λόγους. Πρώτον, ένα ισχυρό σύστημα υγείας παρέχει καλύτερη περίθαλψη στους κατοίκους, αλλά ταυτόχρονα ένα ισχυρό σύστημα υγείας είναι εξασφάλιση για την πρόληψη ασθενειών και επιδημιών. Αυτό το οποίο λοιπόν μας λείπει, αυτό στο οποίο υστερούμε, είναι επενδύσεις στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Και όπως είπα και νωρίτερα, η οικουμενική κάλυψη υγείας και τα ενισχυμένα συστήματα υγείας είναι οι δύο ύψεις του ίδιου νομίσματος. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει και να επενδύσουμε στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Θα είναι εξασφάλιση για μας. Τώρα, πολύ σύντομα για τη μετανάστευση και τη γειτονία. Παρεμπιπτόντως γι' αυτό, νομίζω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της μετανάστευσης, και να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε τα συμπτώματα, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τις ρίζες του προβλήματος. Συγκρούσεις, ε, ένδια, ανεργία, όλα αυτά πυροδοτούν την κατάσταση, έλλειψη πρόσβασης σε παιδεία, σε εκπαίδευση. η απάντηση δεν είναι να παραμελήσουμε την υγεία. Πρέπει να επενδύσουμε καλύτερα σε υγεία και σε εκπαίδευση, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως το αποκαλούμε, και θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε επίπεδο χώρας και επομένως να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα. Επένδυση σε στρατηγικά συστήματα είναι καλύτερη. Ε, το να διαχειριστούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο μετανάστευσης ε, τώρα δεν θα το σταματήσει. Είναι σαν ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλύτερη μακροχρόνια λύση. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική λύση και αυτή νομίζω ότι είναι η απάντηση. Δεν νομίζω όμως ότι θα το σταματήσουμε εάν ε, αμελήσουμε να επενδύσουμε την αντιμετώπιση των αιτίων του προβλήματος και αυτό πρέπει να γίνει στην πηγή. Όσον αφορά τη μικροβιακή εντοχή, ενημερωτικά τα προηγούμενα προγράμματα, σας το είπα ήδη, είχαν κάποια αποτελέσματα και το τελευταίο είναι ότι η υγεία θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πέραν της ιατρικής περίθαλψης. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια πολετομιακή προσέγγιση, όπως είπε και κάποιος ευρωβουλευτής, διότι ε, οι παράγοντες της υγείας ε, μπορεί να είναι εμπορικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, μπορεί να είναι και περιβαλλοντικοί. Το να βρούμε λοιπόν τα αίτια του προβλήματος, ε, να αντιμετωπίσουμε από πού προκύπτει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να έχουμε μια πολυτομεακή προσέγγιση και βάσει και των στόχων ε, της βιώσιμης ανάπτυξης ε, υπάρχει αυτό το αίτημα. Προτείνουμε να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές με χώρες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με πολυτομιακή προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Συγγνώμη αν παρέλειψα κάποιε, αλλά νομίζω ότι απάντησα στι περισσότερε. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι βλέπω γνέφουν ε, καταφατικά οι συνάδελφοι, άρα μάλλον του καλύψατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δόκτωρα Τρέβος και την Σουζάννα Γιακο. Θα έπρεπε να είχα πει ότι η Σουζάννα ήταν επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον έλεγχο των ασθενειών. Τη γνωρίζω από τότε που ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας. Οπότε, σας ευχαριστούμε πολύ, Δόκτωρα Τρέβος, και ελπίζουμε να είμαστε σε επαφή ακόμα. Να έρθουν οι επόμενοι προσκεκλημένοι μας, παρακαλώ, εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάνουμε στους επόμενους εξαίρετους ε, ομιλητές. Είχαμε για τη μετανάστευση πριν, είχαμε από τον ΠΟΙ στη συνέχεια και τώρα θα μιλήσουμε για τα δάση και με την UNEP. Είναι το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων με τον νέο επικεφαλή για τα θέματα των δασών, διαχείριση φυσικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες σε περίπτωση των δασών. Η Χάιντι Χαουτάλα είναι συγγήτρια, αλλά ο κ. Μαρσελέση θα την αντικαταστήσει. Έχουμε μελέτη της Επιτροπής για την κατάσταση στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες του 2016 και πήγαμε στο Καμερούν η επιτροπή μας δηλαδή, μια αντιπροσωπεία της, για να δούμε την κατάσταση εκεί. Και τώρα ετοιμάζουμε έκθεση πρωτοβουλίας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, βάση του 54 και με ιδιαίτερη χαρά έχουμε σήμερα δύο ομιλητές, τον Τιερή Λούκας που είναι επικεφαλής του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον στο γραφείο των Βρυξελών και τη Χατουβαριλίση, η οποία είναι η υπεύθυνη από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Την γνωρίζουμε γιατί είχε προετοιμάσει διάφορα θέματα για την διάσκεψη της αντίσαμπεβα, οπότε την γνωρίζουμε ήδη. Δεν έχουμε το σχέδιο έκθεσης. Θα ακούσουμε τους δύο ειδικού. Θα δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στον κύριο Λούκας και μετά στην κυρία Μαριλίσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάβεν. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ήρθα να σας παρουσιάσω τη θέση του ΟΗΕ και θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάτι που θα συμπληρώσει βέβαια και συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ για το που βρισκόμαστε. Αν φελτιώσετε την βιοπικιλότητα, τότε γίνονται πιο ανθεκτικά τα οικοσυστήματα. Και έτσι αυτά που θα συζητήσουμε τώρα έχουν να κάνουν και με το επόμενο σημείο που έχετε στην μερίσια διάταξη, που είναι το θέμα των αυτόχθονων πληθυσμών. Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή. Έχουμε τη Συμφωνία των Παρισιών και πρέπει να πετύχουμε να είμαστε κάτω από τους δύο βαθμούς. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν κοιτάξετε εδώ το διάγραμμα και ελπίζω να μπορείτε να το διαβάσετε, εάν η τροπική αποψήλωση ήταν μια χώρα, τότε, χώρα, τότε οι εκπομπές της θα ήταν μεγαλύτερες από εκείνες συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν θέλετε να πετύχετε τη Συμφωνία των Παρισιών, να την υλοποιήσετε, μπορείτε να το κάνετε με ή χωρίς τα δάση. Αν το κάνετε με τα δάση, τότε θα είμαστε κάτω από τους δύο βαθμούς της θερμοκρασίας. Θα είναι και πιο φτηνό, γιατί οι επενδύσεις θα αποδώσουν και θα υπάρξει μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις επενδύσεις. Και επίσης θα πετύχετε την υλοποίηση αυτή και πιο γρήγορα. Γιατί βλέπετε ότι θα το πετύχετε πέντε χρόνια νωρίτερα σύμφωνα με το διάγραμμα. Συνεπώς, από σήμερα λέμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ένα 30% της άμβλησης. Αν αρχίσουμε όπως σήμερα. Και οι επενδύσεις βεβαίως θα βοηθήσουν παγκοσμίω. Η Συμφωνία των Παρισίων έχει το άρθρο 5 που ζητάει την προστασία των δασών. Και είναι το μόνο μέτρο άμβλησης των επιπτώσεων που αναφέρεται στη Συμφωνία. Και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πρωταθλήτρια στο άρθρο αυτό 5. Επίσης, οι βιώσιμοι στόχοι αναγνωρίζουν το ρόλο που παίζουν τα δάση. Αλλά τα δάση είναι πολύ σημαντικό για το 25% του πληθυσμού του κόσμου εξαρτάται από τα δάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων, για τη ζωή τους, για οτιδήποτε έχει να κάνει με την ευημερία του κόσμου μιλάμε για θέματα υγείας. Τα δάση βοηθούν την υγεία μας και αυτό το γνωρίζουμε όλο και καλύτερα όσο ο καιρός. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι προσφέρουν καταφύγιο τα δάση σε 300 εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Οπότε κανονικά η ανάπτυξη συνδέεται με την αποψήλωση. Δηλαδή λέμε έχουμε ανάπτυξη ε, κάνουμε αποψήλωση και μετά ενδεχομένω αναδάσωση. Αυτό που εμείς πιστεύουμε όμως στον ΟΗΕ είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή σε όλες τις χώρες και αυτός είναι ο στόχος μας. Να φροντίσουμε δηλαδή ότι έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να περάσουμε κάτω από αυτό το τούνελ. Γιατί αλλιώ ε, περνάει αιώνε. Και δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να περιμένουμε. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία για να ξέρετε τι έχει γίνει ανάμεσα στο 2010 και 2015. Στην Βραζιλία χάθηκε 0,2%, στην Ινδονησία 0,7%, στη Μιαμάρ 1,8% των δασών. Το Ιγκάτσου βρίσκεται ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αργεντινή. Και βλέπετε εδώ ποια είναι η κατάσταση και πώς προχωράει. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει σε πολλά σημεία του κόσμου. Τι χρειαζόμαστε τώρα και ποιο είναι το μήνυμα κλειδί που θέλουμε να σας περάσουμε. Είναι ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε την αποψήλωση από την ανάπτυξη. Δεν περνάμε από την αποψήλωση για να πετύχουμε ανάπτυξη. Και έχουμε τώρα μια πραγματική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Έχουμε τη δήλωση των Παρισίων, όπως είπαμε, τη συμφωνία υπάρχει. Έχουμε την πολιτική άρα βούληση, αλλά έχουμε και το know-how. Ξέρουμε. Έχουμε δουλέψει και στον ΟΗΕ με διάφορα προγράμματα. Ακούσαμε πριν και για την ασφάλεια. Όντως, η ασφάλεια, η υγεία και τα δάση. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι βέβαια και χρήματα. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην πρώτη γραμμή για πολλές ε, δραστηριότητες. 5 δισεκατομμύρια. Η Γερμανία, για παράδειγμα, είναι μεγάλος δωρητής. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε κίνητρα και χρηματοδότηση στις χώρες, ώστε να μην κάνουν αποψήλωση. Αν κατακλείδει, τι χρειαζόμαστε. Τα δάση είναι ουσιώδη, είναι θεμελιώδη προκειμένου να υπάρξει ελπίδα για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισιών. Χρειαζόμαστε επίσης συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν όλοι. Και το τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. 80 χώρες μπορούν να αποφεληθούν από το σχέδιο RED τώρα. Βραζιλία, Ινδονησία. Δεν είναι μόνες, είναι λάθος αν σκεφτόμαστε αυτό. Πρέπει να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Καλό είναι που μιλήσατε για το Καμερούν. Όντω, αυτό πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σαντάλ τώρα. Δεν θα κάνω την παρουσίασή μου. Νομίζω ότι αρκετά PowerPoint είδατε σήμερα. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτά που είπε ο προλαλήσας. Δηλαδή για μας ε, τα δάση είναι ε, πλούσια πηγή, πλουτοπαργωική πηγή, ανέφερε ότι μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, αλλαγή ε, προσφέρουν βιοπικιλότητα, αλλά και εισόδημα σε κάποιους από τους πιο φτωχούς ανθρώπους του κόσμου. Είναι πολύ χρήσιμα τα δάση για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030, αλλά και σχετικά με τη συνένεση που υπάρχει για την ανάπτυξη. Ε, συμβάλλουν στην ειρήνη, στα τρία π, ε, στην ειρήνη, στους ανθρώπους, στον πλανήτη. Τρία π στα αγγλικά. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι ε, υπάρχει πάλι επιβεβαίωση ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράνομη ξυλία ε, και η ε, παράτυπη εκμετάλλευση των δασών. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με καλύτερη διακυβέρνηση και δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων. Για μας για την Επιτροπή Ανάπτυξης, για την έκθεση Επιτροπής ε, σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για τα δάση σε ξένες χώρες. Αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, είναι άλλη μια έκθεση που για μας αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για τα δάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη στο να προσφέρει καλή διακυβέρνηση στον τομέα των δασών και έχουμε μια αναβαρχίδα που ισχύει τα τελευταία 15 χρόνια είναι επιβολή του νόμου, το εμπόριο, η σωστή διαχείριση, το πρόγραμμα δράση, Πρόκειται δηλαδή για ένα ε, ιδιαίτερα διευρυμένο εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, παράνομη ε, παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων από δάση. Ε, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα με την έννοια ότι προσφέρουν τη δυνατότητα να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη της, ε, τις ε, ιδιωτικές κοινωνίες, για όλους όσοι, ασχολούνται με την παράνομη ξυλία και το εμπόριο πρέπει να φτάσουμε στις ρίζες στη ρίζα του προβλήματος και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, αντιμετωπίζει το θέμα της έλλειψης λογοδοσίας και διαφάνειας, την περιορισμένη συμμετοχή, πολύ αδύναμα ε, νομικά συστήματα, ε, την, τα θέματα της εμπορικής συνεργασίας, αλλά και τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων. Αυτό είναι μάλλον συνηθίστο, δηλαδή να υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία να συγκεντρώνει όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια παραδείγματα, ε, θα πούμε και άλλα, αλλά δεν θέλουμε να βαρεθείτε με πάρα πολλά. Αν ε, θέλουμε να, αν θέλετε εσείς να επανέλθετε και να εξετάσουμε και άλλες χώρες, μπορούμε να το κάνουμε αργότερα. Θέλουμε να μιλήσουμε λιγάκι για την Ινδονησία όπου υπάρχει το πρώτο πρόγραμμα ε, αδειοδότησης ε, από τον Νοέμβρη του 2016 και ήδη έχουμε 39.000 αδειοδοτήσεις ε, που προσφέρονται για εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή 1,5 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Ε, δηλαδή 25% των εισαγωγών τροπικής εξηλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα αδειοδότησης να συνεχιστεί. Την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία θα εξετάσουν τον πρώτο ανεξάρτητο έλεγχο αυτού του συστήματος είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, να αναλύσει κανείς όλα αυτά τα θέματα. Ε, το θέμα των αδειοδοτήσεων στην Ινδονησία, αυτό είναι ένα πολύ μακρύ ταξίδι που κάναμε από κοινού με τις αρχές της Ινδονησίας και το ταξίδι αποτελεί το από ε, αλλαγές ουσιαστικές στον τομέα των δασών. Έπρεπε να ελέγξουμε την παράνομη, τις παράνομες ομάδες πίεσης και να τροποποιήσουμε όλο αυτό το σύστημα των αδειοδοτήσεων. Χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο και το ίδιο συνέβη και με την Κάνα, όπου ελπίζουμε ε, τον επόμενο χρόνο οι άδειε να μην προσφέρονται πλέον από την Κάνα. <clears throat> Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να αλλάξει τελείω εκ και το νομικό σύστημα στην Κάνα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικό τομέα μπόρεσε να συζητήσουν τα νομικά θέματα, πώς όλα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται και μάλιστα και με συνενετικό τρόπο. Η θέση που έχουμε εμεί ως εμπορικός εταίρος ε, έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκηθεί πίεση στους εταίρους έτσι ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νομοθετική ε, μεταρρύθμιση. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης ε, το ότι πλέον υπάρχει μία online πλατφόρμα που προσφέρει ε, πληροφορίες για την ξυλία, για τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Αυτή η πλατφόρμα κατασκευάστηκε όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα και ιδιωτικέ εταιρείε. Βλέπουμε ένα σύστημα ε, το οποίο έχει συσταθεί από ε, διάφορους που κατά κανόνα δεν συνεργάζονται. Στις Ονδούρες. Αυτή είναι η τελευταία χώρα που ζήτησε ε, διαπραγματεύσεις ε, και θα ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις σιγά σιγά. Ε, αρχές του καλοκαιριού θα ξεκινήσει η διαπραγματεύση με τις οντούρες. Πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, γιατί είναι μια χώρα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή για την καλή της διακυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλησε να μεταρρυθμίσει τα δάση, τον τομέα αυτό, όχι μόνο για να προσποριστεί χρήματα, αλλά για να έχει και μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς. Είναι το πρώτο πρόγραμμα όπου βλέπουμε οι αυτόχθονες να συμπεριλαμβάνονται στις ε, διαπραγματεύσεις. Εγώ όταν ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με την Ονδούρα, είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι εντυπωσιάστηκα γιατί δεν διαπραγματευόμουν με την κυβέρνηση, αλλά με την κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα, τους αυτόχθονες και άλλες οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών. Και όλοι αυτοί καθόντουσαν μπροστά μου, ε, μπροστά στο βίντεο ε, και τους ρώταγα αν συμφωνούν με την θέση της κυβέρνησης, με τη δική μας θέση και μου έδιναν μια ειλικρινή απάντηση. Όλοι αυτοί ε, πάρα πολύ χρήσιμο. <clears throat> Επίσης, με τις Ονδούρες βλέπουμε την πρώτη προσπάθεια να συμπεριληφθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ομοθεσία ε, για την ε, συνένεση ε, δεν είναι τέλεια η όλη διαδικασία. Δεν θέλουμε βέβαια να ασκήσουμε πίεση, γιατί δεν θέλουμε να φανεί ότι πιέζουμε για ένα νόμο που δεν είναι αρκετά καλός, όμως έχουμε πλέον το χώρο όλα αυτά να συμπεριληφθούν στο σύστημα και να επιτρέπεται στην κυβέρνηση και στην κοινωνία των πολιτών να συζητήσουν αυτό που μακροπρόθεσμα ε, θα είναι ένας καλός νόμος ε, και θα μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από το πρόγραμμα VPA και το σύστημα της αδειοδότησης και άλλες χώρες, το Καμερούν που αναφέρατε, η Δημοκρατία του Κονγκό, όπου υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις ε, η χώρα DRC, η δημοκρατική, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και εκεί έχουμε διαπραγματεύσεις που επανέρχονται η Γκουιάννα και εκεί ε, ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις ε, μέχρι να ε, υπάρξουν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις σε οποίες επιθυμούν να προβούν. Με διάφορες χώρες έχουμε εμπειρίες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ θα μπορούσα να σε ενημερώσω και για άλλες εργασίες που κάνουμε για την αποψήλωση. Αλλά ολοκληρώνουμε και το πρόγραμμα που θα τρέξει μέχρι το 2022, όπου έχουμε ως στόχο να εξορθολογήσουμε όλα αυτά που κάνουμε κάτω από την ε, ε, εμβληματική πρωτοβουλία. Μας λένε ότι ε, δαπανάμε πολύ χρόνο για τα DPA, παρότι όμως είναι ακρογωνιαίος λίτος ε, και όπου υπάρχουν πολλοί άλλοι όπου συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε καλύτερο έλεγχο της εξηλίας, καλύτερο προγραμματισμό των δράσεών μας. Και αυτό το εξετάζουμε και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τη συζητήση με τα κράτη-μέλη τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι βλέπετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόσμο από τότε που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια η εμβληματική πρωτοβουλία. Προφανώς και παραμένουμε δεσμευμένοι στην αντιμετώπιση της λαθροξυλίας, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή συμβάλλει στην αποψήλωση και γνωρίζουμε ότι δεν είναι ε, η μόνη αιτία της αποψήλωσης ε, και οι εξορίξεις ε, και πολλές άλλες παράνομες δραστηριότητες οδηγούν στην αποψήλωση. Φινικέλαιο, καφές και αυτά μεταξύ άλλων είναι αίτια που οδηγούν στην αποψήλωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές έμεσες ενέργειες που οδηγούν στην αποψήλωση, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παρανομίες και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα του νομικού πλαισίου, της σωστής εφαρμογής του νόμου. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα αν θέλουμε να περιορίσουμε την αποψήλωση και προφανώς να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η εμβληματική πρωτοβουλία και τα VPA προσφέρουν πολύ σημαντικούς ε, τρόπους, για το, μάλλον για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ευρύτερο θέμα της αποψήλωσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι ακριβώς έχουμε μάθει τα τελευταία 15 χρόνια. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει δύο ανεξάρτητες μελέτες εμπειρογνωμόνων που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ταιριάζουν και στη δουλειά που θα κάνουμε εμείς στο μέλλον για την αποψήλωση. Ε, πρέπει να σας πω, δεν περιμέναμε αυτές τις μελέτες. Ο Τιερή σας είπε ότι έχουμε μελέτες που μας προσφέρουν πρωτοβουλίες υπό που μας προσφέρουν πληροφορίες υπό τον πρωτοβουλία RED. Και θεωρούμε ότι ε, υπάρχει και η εμπειρία πολλών κρατών που είναι πολύ χρήσιμη, ε, τον δεκαετής εμπειρία, ε, πολύ χρήσιμη, γιατί υπάρχουν πάρκα τα οποία δίδονται για την ξόριξη πετρελαίου και αν συνεχίσουν όλα αυτά θα εξακολουθήσουμε να έχουμε την αποψήλωση και την επιδείνωση της κατάστασης στη γη. Η αποψήλωση είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Αν δούμε τα βασικά αγαθά, τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στην αποψήλωση, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν αντιμετωπίσουμε την αποψήλωση στην ε, αλυσίδα αξίας ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην υπάρξει μετακίνηση ε, σε άλλες μορφές γεωργίας, την γεωργία επιβίωσης. Ως εκ τούτου ε, τα δάση πρέπει να συνδυάζονται και με το περιβάλλον, αλλά και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και εισόδημα για τους ε, πιο φτωχούς λαούς του κόσμου. Να υπάρχει μια ισορροπημένη ε, προσέγγιση οποτεδήποτε εργαστούμε και στο μέλλον για την αποψήλωση. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι έγκυρη λοιπόν η έκθεσή μας, αν και εσείς σκοπεύετε τώρα να καταρτήσετε το τετραετές σχέδιό σας και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι υπάρχει μελέτη που εκπονήθηκε πέρσι και είναι διαθέσιμη από τη Διεύθυνση Πολιτικής που σας δίνει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για το FLEGD και αναφέρεται νομίζω η Γκάνα, η Τανζανία, δεν θυμάμαι ποιες άλλες χώρες και το Καμερούν ε, στην έκθεση εδώ. Η Χάιντι Χάουτολα απουσιάζει, αλλά έχουμε τον κύριο Μαρτσελέση, ο οποίος ε, την αντικαθιστά. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, σήμερα η Χάιντι απουσιάζει, αλλά είναι στο Ελσίνκι. Ε, και επομένω χαίρομαι που την αντικαθιστώ γιατί μπορώ να ε, συμμετείχα μάλλον και στην αποστολή στο Καμερούν στο θέμα της αποψήλωσης και να ξεκινήσω και να πω ευχαριστώ για την παρουσίαση γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ε, ε, τα οποία έχουν προχωρήσει και συμφωνούμε με αυτά που είπατε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη Ηνωμένα Έθνη και χαίρομαι που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για την καταπολέμηση αποψήλωσης, διότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή ε, κλειδί για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Το είπατε κι εσείς, υπάρχει η Συμφωνία των Παρισίων που μας επιτρέπει να θέσουμε τα βάση στο επίκεντρο της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είπατε πολύ καλά. Υπάρχουν ε, το 30% της δυνατότητας μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και 20% των εκπομπών ε, του, αερίου του θερμοκηπίου ε, είναι λόγω των δασών και της αποψήλωσης. Επομένως, αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αποψήλωση, δύσκολα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Συμφωνίας των Παρισίων. Και επίση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θέτε στο επίκεντρο της δράσης τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τα δικαιώματα που έχουν επί της γης, γιατί ε, έτσι θα μπορέσουν να προστατεύσουν τα δάση και να αποφύγουν την αποψήλωση. Κάποιε από τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνονται ενδιαφέρουσε και νομίζω ότι μπορούμε να τις ε, στηρίξουμε και εμεί από πλευράς Επιτροπής. Δέωσα επιμέλεια και κανονισμός για την αντιμετώπιση των αγαθών από τα δάση, ε, επίσης ε, αντιμετώπιση τη αποψήλωση επενδύσεων και ε, χαμηλότερους δασμούς εισαγωγής για αγαθά τα οποία βοηθούν τη βιώσιμη παραγωγή ή και τα κριτήρια της αποψήλωσης ή ε, κριτήρια, κριτήρια βιωσιμότητας. Ε, πιστεύω ότι αυτά είναι τέσσερις προτάσεις που μπορούν να μας βρουν σύμφωνους από πλευράς Επιτροπής Ανάπτυξης. Είναι ουσιαστικά στοιχεία και επιπλέον θεωρώ ότι θα πρέπει να μας πείτε πώς σκοπεύετε να υλοποιήσετε ή πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποψήλωση. Νομίζω ότι εδώ και καιρό το ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το σχέδιο. Καλό θα ήταν να μα δώσετε κάποιε περαιτέρω πληροφορίε. Επίση να σα πω ότι και η Χάιντι ε, προχωρά αυτή τη γνωμοδότηση ίδια πρωτοβουλία για την αποψήλωση και να σα πω ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα περιλαμβάνει. Καταρχά ε, όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένω, συμφωνώ ε, και σε αυτά είδαμε και στην αποστολή στο Καμερούν και έχουμε τα εξή. Θα επικεντρωθούμε καταρχάς στην επέκταση της γεωργίας, ε, την αντιμετώπιση της αποψήλωσης και τι συνέπειες μπορεί να έχει για αυτόχθονες πληθυσμούς. Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά ό,τι έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση της γης, ε, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, ε, διότι η διαφθορά είναι στο επίκεντρο όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αποψήλωση στις χώρες που μας απασχολούν. Να υπενθυμίσω επίσης ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη υλοποίηση του FLEGD και των σε ειδικών προγραμμάτων, γιατί ήταν ένα εργαλείο το οποίο ήταν καινοτόμο μεν, αλλά αν δούμε τι συμβαίνει στο Καμερούν, ε, δεν είναι πανάκια για όλα. Πρέπει λοιπόν να τα ξαναδούμε τα θέματα και να δούμε και πώ υλοποιούνται για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μα. Επίση, πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο όχι τι έχει να κάνει με την αλυσίδα προμηθειών και ε, ε λογικές, λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων, συνέργειες επίσης που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ του RED και του FLEGD, διότι ε, ο καθένας λειτουργεί ξεχωριστά από την πλευρά του, αλλά αυτά τα δύο εργαλεία πρέπει να λειτουργούν από κοινού να μιλήσουμε και για την ε, εγκληματικότητα και τα εγκλήματα των δασών. Ε, όταν αναφερόμαστε στην περιβαλλοντική εγκληματικότητα υπάρχουν πέντε τομείς ε, που περιλαμβάνονται και μεταξύ αυτών πάντα τα δάση και μετά περιβαλλοντική διπλωματία, κλιματική διπλωματία να μπορέσουμε να έχουμε μία μόνη συνεκτική πολιτική για τα θέματα αυτά. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία λοιπόν που θα έχει η έκθεση πρωτοβουλία της Χάιντι Χάουταλα και ε, με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλια και ε, τις παρεμβάσεις των σχεδόν εισηγητών για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και νομίζω ότι πλέον κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο, η Σεσίλ Κέγγι και ο Νόμπερτ Νόιζερ. Ο Νόρμπερτ πρώτα και μετά η Σεσίλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, να ευχαριστήσω τη Χάιντι Χάουταλα για την έκθεσή της. Μιλώ εξ ονόματος ε, του ε, ε σκιώδους μας και θα ήθελα απλώς να προσθέσω τη σύντομη δήλωσή του. Η έκθεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει μια σειρά από σημαντικά νομοθετήματα που στόχο έχουν να προστατεύσουν τις ιδιότητες απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα των δασών ανά τον κόσμο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ολοκλήρωσε ένα φιλόδοξο καθεστώς για την αντιμετώπιση των ορυκτών σε περιοχές συγκρούσης, ε, για να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικές ζημίες και ζημίες λόγω σύγκρουσης. Το 2013 είχαμε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμά ότι μεταξύ του 1990 και του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε περίπου το 1 τρίτο όλων των προϊόντων αποψήλωσης που προέκυψαν σε διάφορες περιοχές. Ε, υπάρχουν μια σειρά από διεθνεί συμφωνίε ε, που έχει προσπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει των οποίων δεσμεύεται να μειώσει αυτέ τι ζημίε ε, και την υποβάθμιση και να έχουν περιορισμό των συνεπειών τη κλιματική αλλαγή και την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Οι διεθνεί συμφωνίε έχουν επισημάνει επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δάση για του αυτόχθονε πληθυσμού και πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στα σχέδια προστασίας. Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή ε, θα μπορέσει να έρθει εγκαίρω ε, και να παρέμβει για να κάνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει για την ανάπτυξη ενό ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την αποψήλωση και τις ζημίε των δασών. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα ρυθμιστικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα αλλάξει η προμήθεια και ε, δεν θα υπάρχουν οικονομικές ε, συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει αποψήλωση και υποβάθμιση των ε, δασών και κατάχρηση από πλευράς ανθρώπου. Ευχαριστώ. Ο Νόρμπερτ λοιπόν μιλούσε εξ ονόματος πιο σκιώδου και τώρα η Σεσίλ Κιέγκε. Ευχαριστώ Λίντα. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς τους προσκεκλημένους μας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε για μια πολύ σημαντική απειλή για τα δάση της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκού από ένα σχέδιο το οποίο θα αναπτυχθεί τοπικό για νέες παραχωρήσεις δασών σε μεγάλη κλίμακα. Περίπου 75 ε, εκατομμύρια εκτάρια δασικών εκτάσεων που μπορεί να είναι μια έκταση δύο φορές της Ιταλίας και αυτό φυσικά θα έχει και καταστροφικές συνέπειες για το κλίμα και φυσικά και τα μέσα διαβίασης των ε, πληθυσμών που ζουν σε περιοχές ε, δασικές. Θα ήθελα να ξέρω αν γνωρίζετε αυτό το σχέδιο ε, και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι διαθέτεται μόχλευση εναντί της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό υπάρχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και το περιβάλλον μέσω συγκεκριμένων ε, μέσων και συμμετέχουν και σε διεθνή βήματα για τις ε, πολιτικές της περιοχές. Ε, τι θέση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον της παρούσας απειλής της άρσης του μορατόριου και τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να πείσουμε την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διατηρήσει το μορατόριου. Ευχαριστώ. Σαντάλ, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις μια απόπειρα να απαντήσεις ε, στα όσα ρώτησε η Σιλκιάνγκε για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αν ξέρεις το θέμα. Ναι. Ήμουνα στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό όταν ε, έγινε η όλη διαδικασία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά λοιπόν το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα με την κυβέρνηση η οποία επιθυμεί να αναστείλει το μορατόριο το οποίο υπάρχει για την ε, παράνομη ε, βιομηχανική υλοτομία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μορατόριο για την ε, παράνομη βιομηχανική υλοτομία, αλλά δεν υπάρχει μορατόριο για την ρασιτεχνική υλοτομία. Και ήδη χρησιμοποιούνται Ω πρόσχημα η ερασιτεχνική υλοτομία και γίνεται στην πραγματικότητα βιομηχανική υλοτομία. Ήδη λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. μου χωρί. Και έχουμε και πρόβλημα και όσον αφορά ε, το πετρέλαιο και τη διερεύνηση για πετρέλαιο που θέλει να, γίνει, να κάνουν σε κάποιες περιοχές. Το θέμα του μορατόριου ετέθη στην ε, πρωτοβουλία για τα δάση και την αρμόδια επιτροπή της Κεντρικής Αφρικής και αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση ε, αυτής της Επιτροπής έχει ανασταλεί διότι πρέπει να τηρήσουν ε, τα όσα έχουν συμφωνήσει με την Επιτροπή αυτή, την ΚΑΦΗ. Ε, υπάρχει ε, μια επιστολή προθέσεων και πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Και υπάρχει και απάντηση από την ΚΑΦΗ ε, στην οποία, με την οποία είναι εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσει να παραμένει το μορατόριο και να συνεχίσει η λειτουργία του και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και με το νέο κώδικα περιδασών για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε και μια συμβουλευτική διαδικασία η οποία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να προχωρά στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε εξωτερικοί παράγοντες και αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, η οποία είναι κυρίαρχη. Αν αποφασίσουν να κάνουν κάποια πράγματα μονομερός, η χρηματοδότηση από πλευράς κάφη δεν θα προχωρήσει. Θα χάσουν λοιπόν τα χρήματα από εκεί, αλλά αν πιστεύουν ότι μέσω αυτών των παραχωρήσεων των δασών θα έχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης για τον προπολογισμό τους, ε, είναι πολύ περιορισμένα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ε, κάναμε αιτήματα, διαβήματα αμέσω. Ε, οι δωρητέ ε, που είναι στη χώρα πιέζουν όσο περισσότερο μπορούν την κυβέρνηση. Δεν χρηματοδοτούμε άμεσα την κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος που προωθεί αυτή την πρόταση χρηματοδοτούμε τη διαχείριση των εθνικών πάρκων. Εάν δεν χρηματοδοτήσουμε αυτά τα εθνικά πάρκα, θα γίνει αποψήλωση των εθνικών πάρκων ή θα καταστρέψουν τεράστιες περιοχές σημαντικής βιοπικιλότητας που είναι πηγές χρηματοδότησης για τα δάση. Ε, αυτή τη στιγμή είναι δίλημα λοιπόν και για μας, διότι αφενός ε, η παρουσία μας και η χρηματοδότησή μας είναι αυτή η οποία προστατεύει τεράστιες εκτάσεις γης. Ε, σίγουρα δεν δίνουμε ή δεν σκοπεύουμε να δώσουμε τίποτα στο Υπουργείο για να κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με το μορατόριο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ε, ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για το FLEGT για να υπάρχει και ένα βήμα διαβούλευση, όπω έλεγα προηγουμένω, το γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τη κοινωνία των πολιτών και τη κυβέρνηση και να του έχουμε όλου γύρω από ένα τραπέζι, είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για το πρόβλημα του μορατόριου. Αυτά λοιπόν είναι όσα γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά πράγματι υπάρχει πρόβλημα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπω να ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, ωραία, ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας, τους ομιλητές μας. Και τον Απρίλιο θα έχουμε την ε, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Okay. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης, που είναι η εφαρμογή του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις τροπολογίες στην έκθεση του κύριου Γκερέρο, που θα ψηφίσουμε αύριο. Είχαμε 210 τροπολογίες και ο συγκητής συμφώνησε για 29 συμβαστικές τροπολογίες. Οπότε μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι συμβαστικές που θα ψηφίσουμε αύριο. Παρακαλώ, κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα θυμόσαστε ότι πρόκειται για έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας και του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας πώς λειτουργήσαν δηλαδή από τότε που εγκρίθηκαν. Όμως από την αρχή η Επιτροπή μας και εγώ ο ίδιος πρότεινα στην Επιτροπή να χωρίσουμε σε τρία διαφορετικά τμήματα την έκθεση. Ένα τμήμα που να αφορά καθαρά την αξιολόγηση της λειτουργίας των μέσων αυτών χρηματοδότησης. Ένα δεύτερο τμήμα που να ασχολείται με τις προσδοκίες που είχαμε, τι περιμέναμε από τα μέσα αυτά μέχρι το τέλος της περίοδου, μέχρι το 2020 δηλαδή, και ένα τρίτο μέρος που να ασχολείται με το τι περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να συμπεριλάβει στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα αρχίσει από το 2021. Στόχος των δύο τελευταίων, του δεύτερου και του τρίτου βήματος, ήταν να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τον Μάιο όταν θα μας παρουσιάσει την πρότασή της για διαπραγματεύσεις, εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο, να το έχει υπόψη της. Όπως είπε και η Πρόεδρος, υποβλήθηκαν 210 τροπολογίες. ετοιμάσαμε 29 συμβιβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν λίγο πολύ τις μισές από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες τροπολογίες που τις δέχομαι, κατά πάσα πιθανότητα και περισσότερες πολιτικές ομάδες, γιατί προσφέρουν κάποια καινοτομία, κάτι νέο στην αρχική έκθεση, την εμπλουτίζουν. εστιάζονται καλύτερα, είναι πιο πλήρης όσον αφορά το περιεχόμενο. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που συνεισέφεραν με τις τροπολογίες τους στην βελτίωση της τελικής έκθεσης. Γενικά μιλώντας πάντως, η έκθεση αυτή έχει κάποια βασικά στοιχεία με τα οποία συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες. Πρώτα απ' όλα, λέμε ότι χρειάζονται κάποιοι μηχανισμοί αξιολόγησης και εποπτείας πιο αποτελεσματικοί των μέσων αυτοχρηματοδότησης, ότι πρέπει να έχουμε καλύτερα δεδομένα στη διάθεσή μας από ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα. Επιμένουμε επίσης και επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ότι το 20% των προγραμμάτων της ανάπτυξης συνεργασίας να αφιερώνονται σε βασικά κοινωνικά προγράμματα όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Δεχτήκαμε επίσης τη θέση σύμφωνα με την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε στη Δημοσιονομική Συμφωνία, αλλά διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσει τηρούνται και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει περισσότερο στην παρακολούθηση ώστε να υπάρχει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Επαναλαμβάνουμε κάτι που συνηθίζει η Επιτροπή μας, ότι θέλουμε συνέπεια στις πολιτικές. Ζητούμε να ενισχυθεί η εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών και με τις τοπικές αρχές, όχι μόνο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων, αλλά και όσον αφορά τον προγραμματισμό τους. Δεχόμαστε επίση όπως έχουμε κάνει και άλλη φορά, τα καταπιστευτικά ταμεία, αλλά υπογραμμίζουμε ότι πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται όταν προσθέτουν κάτι παραπάνω στα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουμε ήδη. Και βέβαια όταν ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, κάνουμε τη σύσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να φτάσει στο 0,7% αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό βάσει χρονοδιαγράμματος και βάσει μια συνεχούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς το χρονοδιάγραμμα αυτό. Λέμε επίσης ότι τα κονδύλια που πηγαίνουν στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους στόχους ή για άλλες δράσεις. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει ένας βαθμός αυτονομίας στην αναπτυξιακή πολιτική μας απέναντι στο εξωτερικό και τις γενικότερες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των οποίων πορευόμαστε προς το μέλλον. Έχω να κάνω και δύο σχόλια για κάποιες τροπολογίες που δεν θα δεχτώ. Και θέλω να εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν δύο τροπολογίες που αναφέρονται στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Δεν είναι ότι διαφωνώ με το περιεχόμενο των τροπολογιών αυτών. Το περιεχόμενο πρέπει να πάει στην ε, σωστή ομάδα Δεν έχει κανένα νόημα μία έκθεση γενικού χαρακτήρα να συμπεριλαμβάνει κάτι για δύο συγκεκριμένες χώρες. Γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα να καθίσουμε να αξιολογήσουμε σε κάθε χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε τι γίνεται. Θέλω να πω ότι στην ομάδα εργασία υπάρχει ο κατάλληλο ε, χώρο Εκεί που εξετάζεται η αξιολόγηση των ε, κονδυλίων αυτών των χρηματοδοτικών αυτών μέσων, να δούμε τι γίνεται και στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Και μια άλλη τροπολογία που μιλάει για μια αναπτυξιακή τράπεζα, μια νέα δομή. Αύριο στην ημερήσια διάταξη στους συντονιστές έχουμε ένα σημείο όπου θα συζητήσουμε γι' αυτό και θα τοποθετηθούμε. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η τροπολογία δεν έχει θέση μέσα σε αυτή την έκθεση. Υπάρχει και τροπολογία 110 όπου ο συγκητής σας είναι υπέρ. Πρόκειται για διόρθωση στοιχείων. Στο πρώτο σημείο λέει ότι ένας από τους τρεις λόγους διακοπής της κοίησης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ένας από τους πέντε λόγους. Άρα πρόκειται καθαρά για στοιχείο. Και γι' αυτό και θέλουμε να ψηφιστεί χωριστά σε δύο τμήματα αυτή η τροπολογία. εξηγώντας ότι ο εισηγητής είναι υπέρ. Δηλαδή ότι η άμβλος είναι μία από τις τρεις κύριες αιτίες μητρικής ε, θνησιμότητας, ενώ είναι μία από τις πέντε αιτίες. Τώρα, κατά τα άλλα. Θέλουμε ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο να μας επιτρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους για να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Είμαστε πεπισμένοι ότι η αναπτυξιακή πολιτική όχι μόνο επιτρέπει να βοηθήσουμε χώρες και τομείς και κοινότητες που τη χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, αλλά συγχρόνως μεταβιβάζει και μία ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία ταυτιζόμαστε. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ήπια δύναμη η οποία θέλει τη συνεργασία, την ε, βοήθεια και αποτελεί έναν ε, σημαντικό παράγοντα στον κόσμο, όχι εξαιτία της ισχύω τη, είτε στρατιωτική, είτε οικονομική, είτε αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει κοινωνικό πρόγραμμα, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δρά δημοκρατικά και με αλληλεγγύη απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αρίκε. Ο Ιγνάθιο Κοράου. Όχι. Α, και εσείς. Ωραία, ο Ιγνάθιο πρώτα. Και μετά Εσκιώδης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Και επίσης θα ήθελα απλά να αναφερθώ σε κάποιες ε, τροπολογίες που έχω καταθέσει και που αναφέρονται στο ότι με αυτά τα εργαλεία έχουμε επιτύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ορισμένα εξ αυτών ε, έχουν βέβαια αποκλίνει λιγάκι από τον αρχικό στόχο της βοήθειας. Ε, πρόκειται για κάποια διαφορετική προβληματική, πρόκειται για τη μετανάστευση, το άσυλο, την εσωτερική ασφάλεια. Νομίζω ότι έχουμε επανειλημμένα μιλήσει για όλα αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες ε, που κατέθεσα, παραδείγματο χάρη τροπολογία υπαριθμών 27. Εκεί αναφέρεται ότι όλο και περισσότερο τα ε, κονδύλια για την ανάπτυξη χρησιμοποιούνται για διαφορετικού στόχου, για τον έλεγχο των συνόρων και για πολιτική για τη μετανάστευση. Η 49 λέει ότι την τελευταία δεκαετία ορισμένε από τι χώρε, όχι περισσότερε οι χώρε, ε, ω εκ τούτου ε, βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την μείωση της φτώχειας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η κατάσταση παραμένει ακόμα πολύ κρίσιμη. Η τροπολογία 52 αναφέρει ότι η κρίση δημιουργεί νέες αναγκαιότητες, ε, νέες μορφές ε, βοήθειας, τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στο πλαίσιο των μηχανισμών των ε, επιτόπιων μηχανισμών, των ad hoc μηχανισμών. Γίνεται αναφορά και στα καταπιστευματικά ταμεία. Η 66, εκεί γίνεται λόγος για το ότι δεν θα πρέπει βέβαια να αλλάξει το θεματολόγιο για την ανάπτυξη. Η 94, εκεί αναφέρεται ότι ε, το Ταμείο για την Ανάπτυξη πολλές φορές ε, βρίσκεται χρεωμένο και στην 96 αναφέρεται ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλα προγράμματα στις χώρες που τρέχουν σχόλια χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αυτά, αυτές είναι οι τροπολογίες που ήθελα να υπογραμμίσω γιατί ήμουνα και εισηγητής του Αφρικανικού Καταπιστηματικού Ταμείου όπου έχουμε ζητήσει επανειλημμένα τη διαφάνεια, την εύκολη πρόσβαση ε, και πολλές φορές έχουμε πει ότι το θέμα της διαχείρισης είναι ε, μη διαφανές. Ε, γι' αυτό λοιπόν θέλω να συζητήσουμε τέτοιου είδους και ελπίζω ότι σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε τώρα τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Ρίκε για την διάθεση που απέδειξε για συμβιβασμούς, συμβαστικές τροπολογίες, κάτι το οποίο μας επέτρεψε να καλύψουμε ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού μηνύματος που θέλουμε να στείλουμε, ελπίζοντα ότι τελικά θα εγκριθεί από όλου και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια. Πολύ θετικό. Γιατί στο κάτω-κάτω έχει να κάνει με χρήματα, έτσι, και το χρειαζόμαστε. Τρία πράγματα θέλω να αναφέρω. Πρώτον, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ότι έχουμε πάρει το σωστό δρόμο όσον αφορά ε, την ε, στήριξη του προπολογισμού. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε κονδύλια ούτε για την ανάπτυξη. Πρέπει να υπάρχει αποδοχή και να δίνουμε το σωστό μήνυμα ως Αναπτυξιακή Επιτροπή και το μήνυμα αυτό βέβαια συνδέεται με τις κυβερνήσεις, έτσι. Γιατί ποιοι είναι οι αποδέκτες. Ο κόσμος, οι δικαιούχοι στις χώρες μέλη ζητούν τέτοιου είδους διακυβέρνηση όπως προτείνουμε κι εμείς. Είναι η σωστή προσέγγιση. Με όλες τις εγγύσεις βέβαια που θέλουμε να έχουμε και που είναι σωστό. Για το θέμα της αναπτυξιακής τράπεζας πιστεύω ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι μια καλή ιδέα. Και αυτό για πολλούς λόγους. Και κυρίως μάλιστα γιατί πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε τις επενδύσεις, αλλά και επιπλέον πώς θα εγγυηθούμε για επενδύσεις σε πιο προβληματικά περιβάλλοντα. Αν το θέλουμε αυτό, αν θέλουμε να υπάρχει αυτή η εγγύηση επενδύσεων, Ποιος θα μπορέσει να την προσφέρει αυτή την εγγύηση καλύτερα από μια τέτοια τράπεζα όταν οι διάφοροι επενδυτές της χώρας τους δεν έχουν έναν τέτοιο συνομιλητή. Είναι καλή ιδέα. Μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να κάνουμε και μια έκθεση πρωτοβουλίας ενδεχομένω. Η ερώτησή μου όμως τον Ρίκη και σε όλους μας είναι εξή η συμφωνία που λέει ότι θα συζητήσουμε για την ε, τράπεζα αυτή την αναπτυξιακή δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται η τροπολογία. Και πρέπει να δούμε πώς συνδέεται με την ε, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν νομίζω, ε, συγγνώμη, επενδύσεων. Αν θέλουμε να ψηφίσουμε την τροπολογία, πρέπει να το ξέρουμε. Αλλιώς όλες οι τροπολογίες θα πρέπει να ε, μην έχουν τίποτα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να αντικατασταθεί ενδεχομένω από την αναπτυξιακή. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει. Πάντως αν παραμείνει η τροπολογία θα μπορούσαμε να δεχτούμε μια προφορική τροπολογία στην αρχή, πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε, που να φερεί το, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και τέλος, να ρωτήσω κάτι τη Λόλα. Και αυτό γιατί υπάρχουν διάφοροι στο ΕΛΚ οι οποίοι τρομάζουν όταν ακούνε τέτοια. Η 110 υπενθυμίζει γεγονότα, λέτε. Και άμα πρόκειται για γεγονότα, εντάξει, γιατί να μην υπερψηφίσουμε. Αν είναι ε, η άμβλωση ένας από τους τρεις ή τους πέντε λόγους ε, θνησιμότητας. Τα άλλα όμως μετά για την αναπαραγωγική υγεία δεν με ικανοποιεί σαν διατύπωση. Θέλω να ξέρω. Γιατί δεν επιθυμίζουμε μια νομική βάση την οποία εγώ δεν γνωρίζω. Οπότε παρακαλώ να με βοηθήσετε με αυτό. Αν ναι, θα είμαι προοδευτικός και δεν θα αντιταθώ. Λόλα, θα το κοιτάξετε για την τράπεζα. Όντως είναι ένα επίμαχο θέμα, γι' αυτό και λέμε ότι θα έπρεπε να γίνει σε βάθος συζήτηση. Λόλα, είσαστε σκιώδης συζητήτρια. Θέλετε να πάρετε το λόγο ή όχι. Όχι, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Ωραία, πού είναι ο καταλογός μου. Σεσίλ Κέγγε. Ευχαριστώ Λίντα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον Ενρίκε για τη δουλειά που έκανε και για το έγγραφο το οποίο μας υπέβαλε πάρα πολύ ενδιαφέρον και αποτέλεσε και λίγο μπούσουλα για τη συζητήση μας. Ε, υπέβαλα κάποιες τροπολογίες ε, για να θέσουμε στο επίκεντρο τη διασπορά σε κάποια κεφάλαια, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε 10 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι είναι από χώρε ε, για τις οποίες προορίζουμε τα κονδύλια της αναπτυξιακής βοήθεια ε, και μαζί έχουν αποκτήσει κοινέ αξίε για την καταπολέμηση τη ένδυα, ε, χάρη και στι προσπάθειέ του. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να του έχουμε και στο επίκεντρο ε, μια πολιτική που πρέπει να του αναγνωρίζει και το ρόλο του. Ε, ένα δεύτερο σημείο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι σημαντικό για το θέμα αυτό, είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία προβλέπουν ε, στενή σχέση μεταξύ των ε, κονδυλίων που δίνονται και των ιδιωτικών κονδυλίων της Διασποράς. Θα μπορούσε να είναι η πιο καινοτόμα πτυχή των μελλοντικών προγραμμάτων μετά το 2020 και μία από τις πιο ασφαλείς οδούς για την καταπολέμηση της φτώχειας δεδομένου ότι η διασπορά μέσω ε, αυτών ε, επενδύουν πολύ σημαντικό ε, ποσό στις χώρες καταγωγής τους μέσω των ε, ε, εμβασμάτων. Επομένως προσπάθησα να συμπεριλάβω και αυτή την πτυχή μέσω τροπολογιών. Το δεύτερο είναι το θέμα του ελέγχου. Εκεί κατέθεσα μια τροπολογία που αφορά την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου. Είδαμε μέσω και των αποστολών παρατήρησης των εκλογών σε ορισμένες περιπτώσεις η οικονομική βοήθεια αποτέλεσε ένα μοχλό βάσει του οποίου οι κυβερνήσεις ε, ε εκμεταλλεύτηκαν ε, την κατάσταση. Επομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εις ε, παρακολούθηση της κατάστασης για να δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια εντός ε, κάποιων χωρών σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και μια τελευταία παρατήρηση, συμφωνώ απολύτως με τον Ερίκε όσον αφορά την όλη συζήτηση για κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα ε, τις για το Ιράν διότι είναι μια συζήτηση η οποία έγινε ε, στην ομάδα εργασία και εκεί υπήρχαν συγκεκριμένε επικρίσεις, εξηγήσαμε ποια ήταν η θέση μας, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ε, το μέσο πρέπει να προχωρήσει μεν, αλλά για τις επόμενες φορές... Ε, Καλό θα ήταν να υπάρξει και μια αντιπαράθεση και μια συζήτηση πριν μπορέσουμε να εγκρίνουμε το μέσο. Ε, αλλά αυτή τη στιγμή ε, το μέσο πρέπει να το στηρίξουμε ε, ξεκινώντας από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Κοινοβούλιο, που είχε ήδη ε, ζητήσει να υπάρχει ένα μέσο για την όλη συζήτηση για το Ιράν. Στηρίζω απολύτως λοιπόν τη θέση του Ερίκε και πιστεύω ότι το έγγραφο το οποίο προέκυψε και μετά από τη συνεργασία με την ομάδα εργασία προσπάθησε να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό λαμβάνοντας υπόψη και ποιε είναι οι επικρίσεις αλλά ε, και κατ' ουσίαν το γεγονός ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το μέσο. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρώτα. Έχω εδώ, Dev Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ, ΕΚΟ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Να μην μακρηγορήσετε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από την DG DEFCO πρώτα, ο εκπρόσωπος και μετά έχουμε και τους εκπροσώπους από τις άλλες γενικές διευθύνσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ε, βλέπουμε με ευνοϊκό μάτι αυτό το σχέδιο έκθεση. Περιλαμβάνει πολύ σημαντικέ παρατηρήσει, οι οποίε μπορούν να αποτελέσουν και τροφή για σκέψη για την προετοιμασία των προτάσεων που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο ε, σε αυτά που αναφέρετε. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό σημείο και η συζήτησή μας πρέπει να προχωρήσει από αυτού. Η διάκριση μεταξύ της δημόσιας βοήθειας για την ανάπτυξη και τι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, πρέπει να δούμε δηλαδή τι σημασία έχουν ε, η ε, πλειονότητα των ε, ε, κονδυλίων για την εξωτερική βοήθεια και πολλές φορές τα ζητάμε για την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και στο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, πάνω από το 80% των κονδυλίων επιλέγονται για την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προετοιμασία του μελλοντικού μας έργου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καλείται να παρέμβει σε πάρα πολλές χώρες. Ε, το μεγαλύτερο τμήμα της βοήθειά της είναι αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά υπάρχουν και κάποια προβλήματα, κάποια ε, περιφερειακά προβλήματα ή κάποιες βιομηχανοποιημένες χώρες ε, που δημιουργούν και τεχνητούς φραγμούς σε κάποιες περιπτώσεις και ε, η πλειονότητα της ε, εξωτερικής βοήθειας ε, πάντα μπορεί να θεωρείται και είναι επιλέξιμη για αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό λοιπόν για τη συζήτησή μας γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Kim Έλλινγκ στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, να συμφωνήσω και εγώ με την πολύ θετική εκτίμηση του Βανσάν, να πω ότι και εμείς ε, βρήκαμε πολύ χρήσιμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες και νομίζω ότι τονίζουν ακόμα σαφέστερα ε, τα σημεία της έκθεσης όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και κυρίως για την προστιθέμενη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και τον ρόλο των ανθρωπιστικών αρχών και βεβαίως ε, και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ ανάπτυξης και αναπτυξιακής βοήθειας. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για τις οποίες ε, θεωρήσαμε ότι ίσως ε, θα μπορούσαμε να σας εκφράσουμε τις ανησυχίες μας με την άδειά σας κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς η τροπολογία 34 που αναφέρεται στην ε, Παγκόσμια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή ανθρωπιστικής βοήθειας για να συμπεριλάβουμε και την ανθεκτικότητα. Νομίζω ότι αυτό έχει ήδη αντιμετωπιστεί και η προτινόμενη προφορική τροπολογία 3 ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί και να είναι σωστή λύση. Η 102 που θέλει να επεκτείνει τον κατάλογο των ανθρωπιστικών αρχών για να συμπεριλάβει και μία αρχή μη παρέμβαση που βεβαίως δεν είναι τμήμα των ε, διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών αρχών. Και μετά η 106 και η 107 που επίσης ε, έχουν μια συμβιβαστική τροπολογία την υπαριθμών 11. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες ε, αν λέμε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις και οι αρχές ε, και θρησκευτικέ οργανώσεις θα πρέπει να λένε τις απόψεις τους και να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις περιστάσεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ιδίω σε οξύες περιπτώσεις σειράξεων, που ίσως θα πρέπει να τονίσουμε την ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής δράσης. Και τέλος, η τροπολογία 192 που θέλει η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια να συνάδουν με τις χώρες δωρητές και τους στόχους και θεωρούμε ότι όλα αυτά δεν είναι απόλυτα συνεπεί για τους βασικούς στόχους της ανθρωπιστικής βοήθειας. Βέβαια αυτά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα ίσονα σημασία σχόλια. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε πάρα πολύ χρήσιμη αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο τελευταίος, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω στο να χαιρετήσω και εγώ αυτό το σχέδιο της έκθεσης. Είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμη η έκθεση αυτή και ε, επίσης και οι συμβαστικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν νομίζω ότι θα προσδώσουν ε, ποιότητα στην έκθεση. Δύο πράγματα να σχολιάσω. Νομίζω τόσο στην έκθεση αλλά και σε κάποιες ε, τροπολογίες τίθεται αυτό το θέμα της αυτονομίας, της αναπτυξιακής πολιτικής, ο κίνδυνος της διάσπασης. Ε, νομίζω ότι εδώ το καλύτερο απ' όλα είναι η συνένεση για την ανάπτυξη, όπου αναγνωρίζεται ο πρωταρχικός στόχος που είναι να μειωθεί η πτώχεια στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Βέβαια να συνδεθεί αυτός ο στόχος και με άλλες ε, προκλήσεις, ε, οι παγκόσμιες προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια, η μετανάστευση και όσον αφορά θέματα ασφάλειας δεν μιλάμε για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μιλάμε και για το αίτημα των ε, χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε να μπορούν οι χώρες χώρες αυτές να προσφέρουν ασφάλεια στους πολίτες τους ή και καλύτερο έλεγχο των ε, συνόρων τους, καλύτερη αντιμετώπιση των ε, λαθροδιακινητών. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση ε, για την ανάπτυξη. Και όλα αυτά σχετίζονται και με την κριτική που ασχείται για το καταπιστευματικό ταμείο. Ε, αναμφισβήτητα, συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το επίπεδο της ενημέρωσης, να υπάρχει έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή ε, δράσεων από το καταπιστευματικό ταμείο. Αλλά σε γενικές γραμμές ε, νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το καταπιστευματικό ταμείο έχει βοηθήσει πολύ όπως στην περίπτωση της ε, κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας, την Κολομβία, τη Συρία, αλλά και γενικότερα για τις μεταναστευτικές ροές. Είναι μια συζήτηση που τρέχει θα υπάρξει έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη άποψη γιατί δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο. Συστήθηκε, ιδρύθηκε για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες. Και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι χαιρετίζουμε αυτά που ελέγχθησαν για το μέλλον ε, του μελλοντικού ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου όπου το σχέδιο της έκθεσης ε, προσπαθεί να προβλέπει κάποια χρήματα για τις βασικές ε, δεσμεύσεις. Επίσης, ε, να προσφέρει και ευελιξία στον αναπτυξιακό ταμείο όσον αφορά τα αποθέματα, αλλά και όσον αφορά και τη χρήση των δεσμευμένων κονδυλίων. Όλα αυτά είναι θετικά που θα συμβάλλουν στη συζήτηση για τη νέα δημοσιονομική προοπτική. Ρίκε, έχετε τίποτα να προσθέσετε γιατί ε, έγιναν κάποια σχόλια. Ναι, βεβαίω. Πολλές από τις παρεμβάσεις που είχαν να κάνουν με συγκεκριμένες τροπολογίες που υποβλήθηκαν έχουν να κάνουν με τη τελική θέση του εισηγητή, τον κατάλογο ψηφοφορία. Όταν το δούνε δεν θα έχουν τόσες ανησυχίες γιατί τώρα εξέφρασαν πολύ κάποιες ε, ανησυχείς για το τι θέλει ο συγητής. Όταν μιλήσαμε για την μη ανάμιξη σαν μια βασική αρχή για την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν παίρνει γιατί δεν πρόκειται για αρχή της ανθρωπιστικής μας δράσης, οπότε δεν θα υπάρχει στην έκθεση. Τώρα για να απαντήσω απευθείας για τον Ιγνάσιο Κορέο. Όταν βλέπει τη θέση για τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες παραμένουν και δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικέ, θα δει ότι ακόμα και αν δεν είναι με την διατύπωση ακριβώς τη δικιά του και το ότι υπήρξε πίεση στα μέσα ώστε να στραφούν προς κάποιες πολιτικές μετανάστευση, ασφάλεια ή το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες, πολλές, λίγες, που τήρησαν. Θέλω να πω ότι θα δείτε ότι στο τέλος η διατύπωση θα ικανοποιήσει στο τέλος όταν θα φτάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Θα δείτε ότι η διατύπωσή μου θα σας ικανοποιεί. Τώρα για την δημοσιονομική στήριξη συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Έγγελ και για την διακυβέρνηση ίσως και να είναι το πιο σημαντικό του budget support. Γιατί σημαίνει ότι απαιτεί και βοηθάς τη χώρα να έχει ένα σύστημα διακυβέρνησης που θα της επιτρέψει να επωφεληθεί από την ευκαιρία που της δίνεις με την χρηματοδότησή σου. Άρα δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι θεσμικό, είναι θέμα αξιών, διακυβέρνησης, δημοκρατικών αρχών και ελέγχου. Τώρα για την τράπεζα. Ειλικρινά πιστεύω ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... αν, ναι, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, να μην προκαταλάβουμε εμείς με τη δικιά μας τη θέση κάτι που θα θέλει να κάνει μετά η Επιτροπή μας, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δικιά μας Επιτροπή Ανάπτυξης. νομίζω ότι πρέπει να παρετεθεί ο συντάκτης από αυτήν την τροπολογία. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και δεν είναι ότι είμαι κατά της πρότασης του Φρανκ, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν λαθασμένο μήνυμα να αποφανθούμε εμείς για κάτι για το οποίο ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να έχει λιτά τα χέρια, ώστε να συζητήσει οι πολιτικές ομάδες μεταξύ τους και να καταλήξει αργότερα. Στη ΣΕΣΥΛ θέλω να πω ότι οι τροπολογίες της για τη διασπορά ήταν πολύ χρήσιμες. Έτσι θα συμπεριλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Φωνή και τη φωνή εκείνων που έφτασαν στα σύνορά μας, στις χώρες μας, ακριβώς γιατί έχουν λίγες ευκαιρίες στις χώρες προέλευσής τους και συνεπώς βλέπουν τα πράγματα με πολύ χρήσιμο τρόπο όσον αφορά την ανάπτυξη και τις πολιτικές που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Τώρα για τα σχόλια της Επιτροπής και εγώ συμφωνώ για το ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να συζητήσουμε τι σημαίνει ο όρος αυτονομία της αναπτυξιακής πολιτικής σε ένα κόσμο που αλλάζει, όπου εξελίσσονται οι ανάγκες, οι διάφοροι παράγοντες. Για παράδειγμα, ήμουν συνεισηγητής έκθεσης της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ε, ασφάλεια έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή πολιτική, γιατί διασφαλίζουν ειρήνη και σταθερότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα κονδύλια για την ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιούνται στην πολιτική σταθεροποίηση των χωρών αυτών που μπορούν να βρούνε άλλες πηγές χρηματοδότησης μέσα από άλλους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ισχύει αυτό και για τα καταπιστευματικά ταμεία. Και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να είναι κανείς απόλυτος, χωρίς λόγο. Και επειδή και εγώ είμαι κάποια ηλικία, Λέω ότι δεν πρέπει κανείς να είναι απόλυτος και πρέπει να υπάρχει ισορροπία για να αντιμετωπιστεί κάθε πρόβλημα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο στην ψηφοφορία θα ζητήσω από την ε, Πρόεδρο πριν την ψηφοφορία να μου επιτρέψει να πω δύο λόγια για να ευχαριστήσω άλλους. Πρόεδρος, βεβαίως και θα σας δώσουμε το λόγο αύριο πάλι. Έχετε κάνει πολλή δουλειά και εσείς μπορείτε να ευχαριστήσετε διάφορους και εμείς ευχαριστούμε εσάς. Μετά, θα ψηφίσουμε αμέσως μετά την συνεδρίαση που έχουμε και εξημένο των θυρών. Και φτάνουμε στο σημείο 8 που έχει να κάνει για την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοκτόνων πληθυσμών στον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γεών. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση έχει να κάνει και με τα δάση που συζητήσαμε πριν και με κάτι που συζητήσαμε τον προηγούμενο μήνα για την Κένια για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για το νερό που βοηθάει τους αυτόχθονες πληθυσμούς εκεί. Οπότε με ιδιαίτερη χαρά Έχουμε τον Φρασίσκο Ασής εδώ, που είναι επί τη ουσίας εισηγητής. Θα δώσω πρώτα το λόγο στη Μαρία Χάμπεχ, που είναι η δικιά μας συντάκτρια γνωματότητας, και μετά στον Φρασίσκο Ασής. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Και βεβαίως, ε, Λίντα, έχεις ε, απόλυτα δίκιο ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία ε, έχει σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα δάση μας ανά τον κόσμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιλήφθηκε αυτού του θέματος και αυτής της ε, έκθεσης και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καλούμεθα να τοποθετηθούμε κάτω από το πρίσμα της ανάπτυξης. Έχουμε Κένια και Ονδούρα που πριν από ένα μήνα αναφέρθηκαν και μας δημιουργούν κάποια ανησυχία. Και αυτά καταδεικνύουν τα παραδείγματα ότι ε, έχουν υπάρξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και νεκροί. Άρα δηλαδή όχι μόνο ανησυχούμε, αλλά έχουμε σοκαριστεί. Και όλα αυτά παρά τις, ε, προ... Ε, υποχρώσεις που αναφέρονται στα έγγραφα. Παραδείγματο χάρη, ε, έχω κατά νου την προσέγγιση, τη διάσταση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Οι άνθρωποι αυτοί πάρα πολύ σπάνια μπορούν να δικαιωθούν Υπάρχει λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, υπάρχει αυτή η έκθεση. Σε γενικές γραμμές ε, κατατέθηκαν 81 τροπολογίες ε, που είναι πολύ λίγο για μια μικρή γνωμοδότηση. Αλλά παρόλα αυτά χάρηκα πάρα πολύ για το γεγονός ε, ότι παρά τις τροπολογίες υπάρχει κάποια γενικά η προσέγγιση και βεβαίως ε, θα προσπαθήσουμε αυτές τις ε, τροπολογίες να τις ε, συγκεντρώσουμε σε συμβαστικές προτάσεις και να λάβουμε υπόψη μας και την άποψη όλων των πολιτικών ομάδων. Να σας πω που επικράτησε ευρεία συνένεση. Πρόκειται για την ιδιοκτησία και για τα έθιμα Πρόκειται επίσης ε, για την αρχή που αφορά ε, στην ε, ενημέρωση. Βλέπω ότι χαμηλώνει και το φως. Κατόπιν συνένεση υπάρχει στην αναγκαιότητα συνεργασίας για ε, το θέμα της δέουσας επιμέλειας. Σε αυτά τα τρία βασικά θέματα επικράτησε ευρεία συνένεση και χάρηκα πάρα πολύ που το ΕΛΚΑ αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας διοικητικός μηχανισμός ε, ενστάσεων ε, συμφωνεί το ΕΛΚ και κυρίως ε, στις ε, περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε προγράμματα αναπτυξιακά που χρηματοδοτούνται από τον ΟΔΙΡ, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας διοικητικός μηχανισμός ενστάσεων διότι υπάρχει και ένας άλλος ένας νομικός δρόμος για τα θύματα να μπορούν δηλαδή τα θύματα το συντομότερο δυνατόν να καταθέσουν μία άτυπη ένσταση. Βεβαίω, η νομική οδό ε, δεν αποκλείεται, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι η έγκαιρη ε, δραστηριοποίηση, δηλαδή να είναι αρκετά χαμηλά το κατόφλι για τα θύματα. Και ακριβώς η περίπτωση της Κένιας κατέδειξε πόσο σημαντικός είναι ο μηχανισμός ε, των ενστάσεων. Θα ήθελα να στηρίξετε τις δικές μου τις τροπολογίες, διότι βασικά το θέμα της ε, αρπαγής γεών και το θέμα των ε, ε, δικαιωμάτων που προκύπτουν από το εθνικό δίκτυο. Αυτό θα ήθελα να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη, κυρίως και όσον αφορά και τις επιπτώσεις του κλίματος στους αυτόχθονες πληθυσμούς. Οι τροπολογίες θα έχουν ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. εβδομάδα αν κριθεί απαραίτητο θα ε, συναντηθούμε με τους σκιώδησηγητές. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδησηγητές και αν χρειαστεί τον Απρίλιο θα ε, ορίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ασής έχει το λόγο. Παρακαλώ. Μην ξεχνάτε το χρόνο, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να φύγουν διερμηνείς. Πολύ καλά, θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι παρόν εδώ στην Επιτροπή σας και χαιρετίζω την κυρία Χόιμπουχ για την ε, σύνοψη που έκανε, εξαιρετική και πραγματικά εκφράζει το πνεύμα της έκθεσης. Ε, αυτό παρουσιάσατε ε, με την παρέμβασή σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Η βασική ιδέα είναι η εξή. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του ανθρώπου. Σε όλο τον κόσμο οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν σοβαρά προβλήματα παραβίασης των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιστορικά προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ε, καταστροφή του πολιτισμού τους, ε, αρχαίων πολιτισμών και σήμερα το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ε, πρόβλημα επιβίωσης, ε, πρόβλημα της γης, ε, της ιδιοκτησίας, την επέκταση των γεωργικών συνόρων σε κάποιες χώρες, έκταση εξορρυκτικής βιομηχανίας σε κάποιες άλλες χώρες, ακατανόητες πολιτικές εναντίον των αυτοχθόνων πληθυσμών σε κάποιες άλλες περιπτώσεις από πλευράς κυβερνήσεων και αυτό δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις για την επιβίωση των αυτοχθόνων πληθυσμών. Ε, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στη Λατινική Αμερική, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις και στην Αφρική και στην Ασία. Ε, Υπάρχει μόνιμος διάλογος με μη κυβερνητικές οργανώσεις που μας παρουσιάζουν ε, ε, φρικτές καταστάσεις και ο προβληματισμός μας και ο λόγος για τον οποίο κατατίθεται αυτή η έκθεση είναι για να προβληματιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για θέματα των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Υπάρχουν πάντα εκπρόσωποι και ενός εκπροσώπων και αυτοχθόνων που ε, αναζητούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσουν τις αιτιάσεις τους ε, τρόπον τεινά είναι ένας χώρος ελπίδας ε, για αυτούς τους ε, ανθρώπους από άλλες υπήρους που μας θεωρούν ως ένα κοινοβούλιο που είναι πάντα διαθέσιμο να συζητήσει τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων. Και αυτό είναι τιμή, αλλά ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς ε, τους ευρωβουλευτές. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσιάσαμε αυτή την έκθεση και ε, ξεκίνησε μία συζήτηση με συμμετοχή όλων των πολιτικών ομάδων. Όλοι συνέβαλαν πολύ ουσιαστικά και η Επιτροπή σας παρουσιάζει πολύ σημαντική συμβολή. Ε, συμφωνώ με τον προσανατολισμό της γνωμοδότησης. Μία παρατήρηση μόνο, κάτι που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Κάποια στιγμή στην γνωμοδότηση υπάρχουν κάποιες επικρίσεις για τη σημασία της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ουσιαστική για κάποιε χώρε, για κάποιε περιοχέ και για κάποιου λαού πιο συγκεκριμένα. Επικρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται αυτοί, ε, ε, ε, αυτά τα κονδύλια της αναπτυξιακής βοήθειας και αυτό δεν είναι προ όφελο ε, των αυτοχθόνων. Αφέθηκατε στο θέμα τη Κένια, υπάρχουν και αντίστοιχα θέματα στη Βραζιλία, σε αρκετέ χώρε τη Λατινική Αμερική. Διαπιστώνουμε ότι ε, σχέδια δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την αναπτυξιακή βοήθεια δεν ε, ευνοούν τα ένομα συμφέροντα των αυτοχθόνων πληθυσμών. Και φυσικά η οικονομική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ερώτημα δεν τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σε άλλο επίπεδο και νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα μηχανισμό εγγυήσεων για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αναπτυξιακή βοήθεια ε, σε κάποιες χώρες. Και τέλος να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε. Ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι μια επιτροπή που αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα ε, για τους αυτόχθονες πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νόησελ θέλει να μιλήσει η Λόλα και ο Ιγνάτσιο. Και οι τρεις λοιπόν θέλουν να μιλήσουν. Πρώτα η Μαρία έχει το λόγο. Παρακαλώ. Πολύ σύντομη θα είμαι, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα οποία πολύ σωστά ελέγχθησαν. Μόνο ένα θέμα θέλω να επισημάνω ότι βεβαίως ε, αυτή η εκδίωξη από τις ΓΕΣ, ε, αυτή έχει σχέση και με τη δική μας τη συμπεριφορά και με τη δική μας την κατανάλωση. Το θίξατε αυτό, είπατε ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να δούμε που ενδεχομένως αυτή η πολιτική είναι αντιπαραγωγική. Και αυτό που λείπει είναι ότι κατά την άποψή μου πρέπει να εξάγουμε και συμπεράσματα, τελικά συμπεράσματα. Εμείς τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε άλλες χώρες, μόνο τον εαυτό μας ε, ε, μπορούμε να αλλάξουμε. Ας πούμε εισαγωγέ, φινικέλεου. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί αν δεν το κάνουμε απλά θα περιοριστούμε σε πανηγυρικούς λόγους. Ε, οι χώρες αυτές που δεν είναι δημοκρατίες όποιο ε, έρχεται σε εμπορικέ σχέσει με τέτοιου είδους χώρες, ε, με την έννοια να αγοράζει παραδείγματο χάνει δικαιώματα λίας, αυτό το πληρώνουν πάντα οι πιο φτωχοί των αυτοκτόνων που δεν μπορούν να συμμετέχουν, που ε, δεν μπορούν να βρίσκονται στο τραπέζι των ε, διαπραγματεύσεων. Άρα μόνο η μία ομάδα πλουτίζει και η άλλη γίνεται όλο και πιο φτωχή. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί με ποιες ε, χώρες μπορούμε να συνάπτουμε συμβάσεις και με ποιες χώρες είναι σαπές ότι τα χρήματα αυτά ε, δεν φτάνουν στους πολίτες αλλά στις τσέπες των λίγων. Αυτό πρέπει να το πούμε με απόλυτη σαφήνεια. Δηλαδή η έλλειψη της ε, συμμετοχής των αυτοχθόνων στις αποφάσεις αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η Λόλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ε, είμαι πολύ σύντομη. Ήθελα όμως να ευχαριστήσω τη Μαρία για το εξαιρετικό κείμενο που μας παρουσίασε και χαίρομαι που είναι εδώ και ε, σύντροφος Ασής για να του το πω και του ιδίου. Πραγματικά μας ανησυχούν πολύ οι συνέπειες εξωτερικής μας πολιτικής και θεωρούμε ότι ε, η αρπαγή γεών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει η γη να παραμένει στους αυτόχθονους πληθυσμούς για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά αυτά που έλεγε ο κύριος Ασής ε, και εμεί ανησυχούμε πάρα πολύ για το τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια ε, και να υπάρχει μια σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα και ορισμένες φορές ε, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθών πληθυσμών. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί ε, και να φροντίσουμε ότι αυτή η βοήθεια να δίνεται ε, στους αυτόχθονες πληθυσμούς και να έχουν και συμβουλευτικό ρόλο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε ότι παραβιάζεται το δικαίωμα για διαβούλευση και με αυτούς τους πληθυσμούς. Επίσης, ε, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η αρπαγή γεών στις συμφωνίες που κάνουμε σε εμπορικό επίπεδο και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτές τις αγορές γεών να έχουν και κάποιες μορφές κυρώσεων, γιατί αν δεν υπάρχουν κυρώσεις ε, πάντα θα επιθυμούν περισσότερα. Και πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την αποτελεσματικότητα κάποιων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα, όπω για παράδειγμα στι εθελοντικέ συμφωνίε εταιρική σχέση, το FLEGT και το RED SIN, και να υπενθυμίσουμε ότι από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση εμεί έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την τεχνική και την οικονομική βοήθεια σε αυτά τα μέσα για να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση των δασών. Χρειαζόμαστε επίση, ε, κατά την άποψή μα, και ένα νέο σχέδιο δράση για την αποψήλωση και το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων στη γη αυτών των ε, κοινοτήτων η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώσουν πρέπει να εγκαιάται προστασία σε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα ε, για τα συστήματα των δασών και για τις κοινότητες των περιοχών των δασών και να μην υπάρχει καμία δυνατότητα αποψήλωσης και να συμφωνήσω με τη συνάδελφο Νόιχελ, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα μοντέλα κατανάλωσης. Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο και συνεχίσουμε να ζητάμε κάποια προϊόντα τα οποία προκαλούν αυτά τα προβλήματα, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Λόλα, ο Ιγνάτσιο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Καταρχάς να συγχαρώ και τη Μαρία ε, για την γνωμοδότηση, αλλά και τον Φρανθίσκο Ασής για την ε, έκθεση ε, που είναι από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι τροπολογίες που κατέθεσα κυρίως είναι οι 35 και 63, στις οποίες κάνω συγκεκριμένα μέτρα για να μειώσουμε την αρπαγή γεών και για να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι στις ε, περιοχές των αυτοχθόνων πληθυσμών σε θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμένων. Στην 35 προβλέπεται ένα δημόσιο μητρό για τις ε, περιοχές που κατόχουν αυτέχθονες πληθυσμοί και να είναι γνωστό και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και στην 63 ζητώ μέτρα διαφάνειας από πλευράς εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρέωση να δίνουν πλήρεις πληροφορίες για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με εξορρεκτικές βιομηχανίες ή κάποιε τις αναπτυξιακές ε, δραστηριότητες. Και φυσικά οι πληροφορίες αυτές ε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις ε, διαδικασίες με την κατάσταση και τα εναλλακτικά μέτρα. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα ακούστηκαν προηγουμένως και από τη Λόλα και τη Μαρία και Νομίζω ότι υπάρχει και ένα ηθικό σκέλος στα όσα συζητάμε ε, και στις συνέπειες που έχουν ανά τον κόσμο. Και ελπίζουμε ότι με αυτή την έκθεση και με τη γνωμοδότησή μας να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για ένα μοντέλο που δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. πολύ σύντομα, μόνο αν έχετε κάτι να προσθέσετε, γιατί έχουμε πέντε λεπτά ακόμα ε, διερμηνία και μετά θα πρέπει να σταματήσουμε. Η Γενική Διεύθυνση Να αποτύσω φόρο τιμής σε αυτή την εξαιρετική δουλειά. Πράγματι, είναι δουλειά εις βάθος που επικεντρώνεται σε βασικούς ε, στόχους τα δικαιώματα των ανθρώπων που αφορά η αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε και στη δήλωση και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε προς την πλήρη εφαρμογή που δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Η Κένια είναι μια άλλη περίπτωση στην οποία συζητούμε. Υπάρχει και η δολοφονία ενός ακτιβιστή στο φράγμα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα μαζί. Και το γεγονός ότι ε, σκέφτεστε και ένα μηχανισμό υποβολής ενστάσεων, ε, πρόσβαση σε μέτρα κλπ ε, νομίζω ότι πραγματικά θα προβληθεί, ιδιαίτερα θα είναι μεγάλη προβολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ε, είμαστε μια ισχυρή ε, ένωση με ισχυρή στάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πρέπει να δούμε και τι κάνει ο ιδιωτικό τομέα και να φροντίσουμε να είμαστε καλύτεροι ε, στην ανάπτυξη προ τη σωστή κατεύθυνση για ένα καλύτερο κόσμο. Ευχαριστώ. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, μόνο αν έχετε κάτι να πείτε τίποτα να προσθέσετε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία, έχεις ένα λεπτό. Ε, δεν θέλω και εγώ να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με όλα όσα λέχτησαν εδώ και νομίζω ότι τελικά θα έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Η καταληκτική ημερομηνία για τις, μάλλον ε, στις 24 Απριλίου θα γίνει ψηφορία. Δεν υπάρχει καταληκτική Μάλλον έχει περάσει η καταληκτική ημερομηνία για τροπολογία. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Αύριο το πρωί σε νέα οι συντονιστές και 10 και μισή ε, η ψηφοφορία. Ευχαριστώ τους διερμηνείς για τα επιπρόσθετα λεπτά που μας δώσανε, λέει η Πρόεδρος.